Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε σιγά σιγά. Εγώ θα δώσω τον λόγο και θα φύγω. θα δώσω τον λόγο στον κύριο Κλάιν και θα φύγω. Μ' ακούτε. Ένα, δύο. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και εξ ονόματο 30 εκατομμυρίων ασθενωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εφέκτο, ένα ιατρικό προϊόν, εδώ και 12 χρόνια ε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει γιατί ε, υπάρχει μια αποτυχία εδώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι είναι αυτό το εφέκτο. Είναι ένα μικρό πλαστικό ιατρικό βοήθημα ε, για τους ασθηματικούς, βοήθημα εισπνοής και αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς καθήμενος όρθιος εξαπλωμένος. Είναι η μόνη ε, βοήθεια εισπνοής που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει σε κατάκληση και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα ασφαλείας για τους ασθηματικούς γιατί 70-80% όλων των κρίσεων άσματος συμβαίνουν τη νύχτα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ε, κυκλοφορεί αυτό το προϊόν. Συνήθως τα βοηθήματα εισπνοή έχουν σχήμα γάμα και αυτό δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς ξαπλωμένος. Ε, το πολύ γνωστό Ινστιτούτο Φράουνχοφ έχει κάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη και τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρησιμοποιώ και εγώ αυτό το προϊόν και 30.000 άλλοι από το 1992 τη νύχτα ξαπλωμένο και χαίρο άκρα υγεία. Επίση, επίσης ε, όρθιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανεί και καθήμενο. Τώρα θα σας το ε, ε, επιδείξω. Έχω πάντα το σπρέι για το άσθημα μαζί μου και χρησιμοποιώ έτσι αυτό το μηχάνημα. Δεν είναι ντόπινγκ αυτό. Μην νομίζετε ότι το παρίστηκα τώρα. Ε, και αυτό το σύστημα εφέκτο λειτουργεί θαυμάσια, όχι μόνο σε κατάκληση. Από τότε που χρησιμοποιώ το προϊόν δεν είχα ποτέ κρίση ώστε να πάω στο νοσοκομείο, ούτε σοβαρή. Και αυτό σημαίνει ότι εξοικονομούνται πολλοί πόροι για τα ταμεία. Ε, επίσης ε, και σε φάρμακα. Έχουμε υπολογίσει ότι μέχρι τώρα από το γεγονός ότι δεν κυκλοφορεί αυτό το προϊόν, τα ευρωπαϊκά ταμεία ε, νοσηλείας έχουν χάσει 50 δισεκατομμύρια ευρώ προς μεγάλο όφελος της φαρμακοβιομηχανίας. Και σύμφωνα με την οδηγία της Ένωσης είναι ε, ε, ιατρικό προϊόν της τάξης 1, ε, της κατηγορίας 1, αλλά δεν είναι φάρμακο σε καμία περίπτωση. Φέρει σήμα CE και το κρατήδιο Σαξονία Άχαλ στη Γερμανία το έχει ελέγξει, επιτρέπει την κυκλοφορία. Παρόλα αυτά το αντικρούει αυτό ε, το κρατήδιο της Βαβαρίας που δεν είναι και αρμόδιο να απαγορεύσει την κυκλοφορία του προϊόντος και αναφέρει κάτι αφηρημένους κινδύνους που ενδεχομένως να ενέχονται με το προϊόν ποτέ δεν έχουν αποδειχτεί αυτοί. Το 1997 αυτό ε, οδήγησε σε μια προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι που ε, υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είχε ρυθμίσει αυτό, λέω θα είχε ρυθμίσει σε υποθετικό λόγο γιατί μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει. Τι είναι λοιπόν αυτή η ακρόαση. Γιατί η Κομισιόν δεν έχει κάνει ε, καμία διαδικασία για ε, ασφαλιστικά μέτρα, ασφαλιστική ρήτρα, παρόλο αυτό προτείνεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από μία δεκαετία επικαλούνται οι αρχές κάτι αφηρημένους κινδύνους ε, και ε, αφαίρετα απαγορεύουν την κυκλοφορία ενός προϊόντος που εμπίπτει στην οδηγία 9342 ΕΟΚ και ως ιατρικό προϊόν της κατηγορίας 1. Είναι σε κοφαντίες όλα αυτά που λέγουν και ε, θέλουν να αποτρέψουν ε, η κυκλοφορία του προϊόντος. Ε, ένα κράτος μέλος ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια και τυφλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ακολούθησε ε, για ε, ιδιωτελείς σκοπούς κάποιων εταιριών. Όλοι το λένε, γιατροί, ανεξάρτητοι, βιβλιογραφία, επιστημονική, κλινικά δεδομένα, ότι είναι πάρα πολύ ασφαλές το προϊόν. Πάνω από 200 εκατομμύρια χρήσεις έχουν γίνει από 30.000 ασματικούς από το 1996 και ουδέποτε εμφανίστηκε ενέργεια ή αρνητικό συμβάν που να ε, έχει δηλωθεί ε, στην υποχρεωτική κοινοποίηση. Μα πώς μπορεί ένα προϊόν να είναι τόσο επικίνδυνο που χρησιμοποιείται 14 χρόνια σε πάνω από 200 εκατομμύρια φορές και δεν έχει προκαλέσει τίποτα. Είναι πάρα πολύ ασφαλής αυτή η χρήση και το ιστορικό. Το λένε και τα ταμεία αυτό. Παρόλα αυτά απαιτούν νέε δοκιμέ πριν κυκλοφορήσει στην αγορά. Τα γνωρίζει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ε, δεν αντιδρά και ε, είναι μια ε, ολιγορία συνειδητή. Θα μπορούσαν να είχαν λυθεί όλα αυτά από το 1998 και το αργότερο το 2005 βάσει μιας διαδικασίας που προβλέπεται, αλλά δεν έχει γίνει. Αγαπητέ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Νομική Επιτροπή έχει γνωμοδοτήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίτηδες ολιγορεί εδώ και 10 χρόνια. Είναι σκάνδαλο. Απίστευτο. Να σας πω και τι έγραφε στις 22 Φεβρουαρίου του 2007 στο κράτος μέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι Τώρα θα προχωρήσει στην κινητοποίηση αυτές τις διαδικασίες από το 1997 εκρεμή και θα το κάνει τώρα 10 χρόνια μετά. Μα γιατί 10 χρόνια μετά αφού είναι λέει τόσο επικίνδυνο το προϊόν. Δεν είναι αυτά τα πράγματα παράλογα. Το Φλεβάρι του 2010 το Διοικητικό Δικαστήριο του Μονάχου παραπέμπει σε αυτή την επίσημη επιστολή της Κομισιόν και ε, προχωρεί ένα προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ. Και αυτό χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα για να αντικρουστεί η ε, προσφυγή μας. Εμείς όμως καθόλου τη διαδικασία δεν γνωρίζαμε καθόλου ότι υπήρχε αυτή η επιστολή το 2010. Είχαμε ζητήσει όμως, είχαμε απαιτήσει να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα και τότε μάθαμε ότι υπάρχει αυτό το έγγραφο. Μέχρι τότε υποτιθέμενη ανάλυση της Κομισιόν του 2007 έλεγε ότι δεν πρόκειται να ε, γίνει η διαδικασία αυτή ρήτρα ασφαλείας αλλά εμείς διαμαρτυρηθήκαμε γιατί θεωρήσαμε ότι μας εξαπάτησαν. Το 2007 το Δεκέμβριο ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής Χάιντ Σούρεκ είπε το εξή και παραθέτω. Με βάση τη διαδικασία του 1907 γνωρίζετε ότι δεν δόθηκε συνέχεια και σας έχουμε δώσει όλες τις πληροφορίες. Αν θεωρείτε ότι πρέπει να ακολουθήσετε τη δικαστική οδό, όπως επανειλημμένα αναφέρετε, ή και σε εσά να το αποφασίσετε προφανώς. Παρακαλώ, πώς είπατε, δύο επίσημες γνωμοδοτήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής τελείως αντικρουόμενος για μια διαδικασία υποχρεωτική εδώ και 12 χρόνια. Εμείς ζητούμε να αρθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Βαβαρία και αυτό το απέτρεψαν και το θεώρησαν ε, ε, αντίθετο προς την κείμενη νομοθεσία με ένα προδικαστικό ερώτημα. Κάθε μήνα καθυστέρηση καταστρέφει 300 εκατομμύρια ευρώ στα ευρωπαϊκά ταμεία και ε, επιβαρύνει και καταστρέφει την υγεία των ασθηματικών με υπερβολικές δόσεις και άλλους κινδύνους από φάρμακα που είναι πιο επικίνδυνα από το εφέκτο. Έτσι λοιπόν δεν καταλαβαίνω, ενώ τόσο σαφή τα πράγματα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αποποιηθεί τι ευθύνε τη. Είναι πραγματικά ανεύθυνο αυτό. Και αυτό παρακαλούμε την Επιτροπή σας να συστήσει ε, Επιτροπή εξεταστική έτσι ώστε να διορθωθούν και να ε, διελευκανθούν όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 30 εκατομμύρια σημητικοί δεν έχουν πολιτικό κόμμα και χρειάζονται επιγόντως την υποστήριξή σας. Όπως και οι ασφαλισμένοι, οι ασθενείς και ε, εμείς ε, ως κατασκευαστής. Είναι στη διάθεσή σας και ο δικηγόρος μας, Δόκτωρ Σνάιντερ Αντέα Μένσα. 30 εκατομμύρια σημαντικοί και υποφαινόμενο σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας και την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που αρχίσατε με το θέμα αυτό το απόγευμα. Η Κομισιόν δεν αμφισβητεί ότι το αντικείμενο που εφεύρε ο αναφέρον μπορεί να κάνει εξοικονόμηση κόστους στα ιατρικά για τον ασθενή και για τα ταμεία. Η ευθύνη όμως της Κομισιόν είναι όλες, όλα τα ιατρικά σκευάσματα που κυκλοφορούν στην Ένωση να είναι ασφαλή. Και όπως είπε ο κύριος Κλάιν, τα ιατρικές ε, συσκευές συσκευάσματα διέπονται από την οδηγία του 1993. Αυτή έχει επικαιροποιηθεί πολλές φορές και αυτή τη στιγμή ακόμα βρίσκεται πάλι υπό αναθεώρηση. Ιδιαίτερα με την πρόταση 2011 οι ιατρικές ε, συσκευές σε αντίθεση με τα ιατρικά συσκευάσματα δεν χρειάζονται έγκριση εκ των προτέρων, δεν χρειάζεται να έχουν εγκριθεί από μια κεντρική αρχή, αλλά υπόκεινται σε πιστοποίηση. Και η μορφή πιστοποίησης εξαρτάται από το αν το συγκεκριμένο συσκευή είναι υψηλού ή χαμηλού κινδύνου. Αυτή η συσκευή που εφεύρε ο αναφέρον είναι χαμηλού κινδύνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πιστοποιηθεί ως ασφαλής από τον ίδιο τον παραγωγό, χωρίς παρέμβαση ενός τρίτου, μιας τρίτης αρχής. Ωστόσο, για να μπει απάνω η μάρκα CE, που σημαίνει ότι συμφωνεί με την οδηγία και επιτρέπεται να κυκλοφορήσει ελεύθερα σε όλη την Ένωση, ο παρακατασκευαστής πρέπει να κάνει ένα τεχνικό ντοσχέ με στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλές. Και στο σημείο αυτό έχουμε τις διαφορές μας με τον αναφέροντα. Κατά τη γνώμη της Κομισιόν, ο αναφέροντας δεν κατάφερε να αποδείξει στις γερμανικές αρχές ότι το προϊόν είναι ασφαλές. Ο τεχνικός φάκελος δεν ολοκληρώθηκε. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, ο αναφέρον και ο κατασκευαστής δεν πληρούν τους όρους που θα επέτρεπαν στο προϊόν να κυκλοφορήσει στην αγορά ελεύθερα. Υπάρχουν δύο σημεία εδώ της οδηγίας 9342, το άρθρο 8 σε θέματα ασφάλειας και το άρθρο 18 και τα δύο αυτά άρθρα επιτρέπουν σε εθνικές αρχές να απαγορεύσουν ένα προϊόν. Το άρθρο 8 είναι η είναι ο όρος, η διαδικασία μάλλον για την ασφάλεια. Ένα προϊόν που είναι ήδη στην αγορά, αν για κάποιο λόγο κριθεί από μια εθνική αρχή επικίνδυνο, είτε λόγω ενός ελαιτώματος στην κατασκευή, ή γιατί υπάρχουν νέα επιστημονικά δεδομένα υπέρ του κινδύνου, και με βάση αυτό το άρθρο οι γερμανικές αρχές πρώτον κοινοποίησαν στην Κομισιόν την πρόθεσή τους να απαγορεύσουν το προϊόν του αναφέροντα. Το 1997. Η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε διότι παρόλα τα στοιχεία που είχε τότε η Κομισιόν συν μια επιστολή από τον κατασκευαστή στις γερμανικές αρχές ο παραγωγός, ο κατασκευαστής μάλλον, συμφώνησε να το αποσύρει από την αγορά και δήλωσε ότι προτίθεται να ολοκληρώσει τον επιστημονικό φάκελο. Άρα για μας δεν υπήρχε πιθανότητα το προϊόν αυτό να ξαναεφανιστεί στην αγορά. Ή να αφισβητηθεί η να η απαγορευση Και αυτό εννοούσε και ο κατασκευαστής. Αυτό βγαίνει από μια επιστολή που έστειλε πολύ αργότερα στην Κομισιόν. Το Μάιο συγγνώμη, το 2007. Ξανακούσαμε για το προϊόν αυτό τον Αύγουστο του 2006 όπου αναφέρον ανάφερε στην Κομισιόν ότι κυκλοφορεί το προϊόν στην αγορά με άλλο όνομα και από άλλον κατασκευαστή και ξαναπαγορεύτηκε στην αγορά από τις γερμανικές αρχές. Η Κομισιόν κοίταξε λεπτομεριακά το φάκελο και εδώ καταλήξαμε στο άρθρο 18 που λέει εθνικές αρχές, εδώ η Γερμανία, θα πρέπει να λάβει μέτρα να απαγορεύσει την κυκλοφορία ενός προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με την οδηγία. Οι γερμανικές αρχές θεώρησαν και η Κομισιόν συμφωνεί ότι το προϊόν αυτό δεν είναι σύμμορφο με την οδηγία γιατί δεν υπήρχαν όλα τα δεδομένα από τη μεριά του κατασκευαστή για να αποδείξει ότι είναι ασφαλές. Είναι μια λεπτή διάκριση μεταξύ ενός προϊόντος που δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλές και ενός που έχει αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνο. Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι γερμανικές αρχές σωστά χειρίστηκαν το θέμα αυτό στη δεύτερη περίπτωση. Με βάση δηλαδή το άρθρο 18 ξέρουμε ο Ανεφέρον προσέφυγε στα γερμανικά δικαστήρια είδαμε την απόφαση του ε, βαρικού Διοικητικού Δικαστηρίου του Φεβρουαρίου φέτος ο αναφέρον μπορεί να κάνει έφεση αν θέλει η Κομισιόν δεν έδωσε καμία συμβολή για προδικαστική απόφαση του δικαστηρίου αντίθετα με αυτό που μας είπε ο αναφέρον την απόφαση αυτή την πήρε μόνο του το δικαστήριο η περίπτωση είναι αρκετά σαφής μπορούσε να αποφασίσει χωρίς να χρειάζεται να αναφερθεί στο Ευρωδικαστήριο. Επαναλαμβάνω, ε, έφεση μπορεί να ασκηθεί. Βέβαια, έχει και άλλη λύση ο αναφέρον να δώσει τις αποδείξεις που ζήτησαν οι γερμανικές αρχές μεταξύ του Αυγούστου του 2006 και του Ιανουαρίου του 2008 η Κομισιόν κανόνισε συναντήσεις μεταξύ του αναφέροντα του κατασκευαστή και των γερμανικών αρχών και δόθηκαν ε, συμβουλές λεπτομεριακές στον αναφέροντα τι είδο στοιχεία απαιτούνται για να συμπληρωθεί ο φάκελος με βάση τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή αρκούν συγκεκριμένα δεδομένα που θα στήχιζαν περίπου 30 με 40 χιλιάδες ευρώ στον κατασκευαστή και μερικά φαρμακοκινητικά τεστ σε ασθενεί, αν υπάρχουν ασθενεί που χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Αυτό δεν είναι δύσκολο να γίνει, μπορεί να τα βρείτε στοιχεία αυτά. Η Κομισιόν ε, ε, ε έκανε ό,τι μπορούσε να φέρει σε επαφή τον αναφέροντα με τις γερμανικές αρχές. Και το κάναμε διότι θεωρούμε ότι είναι μια μικρή επιχείρηση, μπορεί να έχει δυσκολία στο να καταλάβει τις υποχρεώσεις που έχει οι γερμανικές αρχές σωστά ερμήνευσαν τον νόμο, η Σάξεν Ανχαλτ που αρχικά δέχτηκε το προϊόν δεν άλλαξε τη θέση της. Συμφωνεί με τις βαβαρικές αρχές να μην είναι στο εμπόριο το προϊόν αυτό. Και αυτή είναι και η θέση της ε, Ομοσπονδιακής ε, Υπηρεσίας για στη Γερμανία ενώ φαρμάκου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Πρέπει να μπει λίγο τάξη στη συζήτηση για να μην έχουμε πάλι καθυστέρηση. Για να έχουμε παρουσία της Κομισιόν μέχρι να κλείσει το θέμα. κύριος Γιάρ, παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η επικεφαλίδα της ε, αναφοράς εδώ ήταν κύλιμη, Με σκοτώνει σιγά σιγά. Εγώ δεν είμαι νομικός. Βέβαια η νομική επιτροπή θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένως οι εθνικές αρχές, πώς να το πω, ασχολούσα μια στρατηγική άρνηση ε, του δικαίου και αυτό δεν είναι σωστό. Με προβληματίζουν εδώ δύο ερωτηματικά. Γίνεται λόγος για το άρθρο 8 και το άρθρο 18. Ο αναφερόμενος το 97 βρήκε ένα νέο πρωτιόν, ένα νέο βοήθημα ιατρικό, κυκλοφόρησε στην αγορά. Εγκρίθηκε από ένα Ομόσπονδο κρατήδιο, ένα άλλο το απαγόρευσε και εδώ μπαίνει μια διαδικασία ασφαλιστική ρήτρα η οποία δεν έχει τελειώσει ή μήπω έχει τελειώσει. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή πραγματικά. Για την ασφαλιστική ρήτρα ενημέρωσαν τον αναφερόμενο ότι ολοκληρώθηκε αυτό. Γιατί το πρόβλημα ποιο ήταν στα γερμανικά δικαστήρια. Δεν μπορεί να βρει το δίκιο του άνθρωπος αν δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο τη διαδικασία. Κάθε πολίτης και επιχειρηματίας έχει δικαίωμα στην ενημέρωση και έχει δικαίωμα στο να γνωρίζει τις αποφάσεις και να λαμβάνονται αποφάσεις, γιατί αυτό είναι εδώ το χειρότερο. Είναι η, η, η έλλειψη αποφάσεων. Γιατί ακόμα και μια κακή απόφαση, απόφαση είναι. Αν ο άλλος αρνείται να αποφασίσει, περιμένω εγώ στην άκρη να δω πότε θα βγει απόφαση και δεν μπορώ να διευκρινίσω την κατάσταση. Και αυτό για μένα είναι το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή την αναφορά. Η μη απόφαση. Και τολμώ να αφισβητήσω ότι αυτή η διάρκεια με όρους κράτους δικαίου είναι ανεύθυνη. Λέω. Δηλαδή αφισβητώ την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το αίσθημα ευθύνης και ρωτώ, αποφασίσατε, δεν αποφασίσατε, ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να ξέρει και τι απόφαση πήρατε. Και αυτή είναι για προσωπική μου άποψη. Θα πρέπει να εκφράσουμε έντονοτατα τη δυσφορία μας. Αρχίσαμε το συζητούμε σήμερα το πρωί. Ό,τι και να γίνει, αυτός που ε, ζητάει κάτι και κάνει μια αναφορά έχει δικαίωμα όχι μόνο στην πληροφόρηση αλλά και στην απόφαση. Ο κύριος Χέφνερ, αυτό είναι πολύ καλό παράδειγμα γιατί έχουμε Επιτροπή Αναφορών και γιατί χρειαζόμαστε το δικαίωμα της αναφοράς. Δεν επιτρέπεται οι προπαίοι πολίτες να παραμένουν χωρίς κανένα δικαίωμα. Έχουμε σαφείς νόμους, από ό,τι φαίνεται αυτοί δεν τηρούνται πάντα όμως. Και καταφεύγει στα δικαστήρια, αλλά αυτή τη φορά δεν μπορεί να πάει ούτε στα δικαστήρια ο αναφερόμενο, διότι είδατε τι έπαθε. 13 χρόνια τον έχουν στο περίμενε. Ο ίδιο έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνία είναι πολύ σημαντικό. Είναι σε εμπλοκή, δεν μπορεί να δράσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να αποφασίσει αν αποφάσιζε θετικά θα συνέχιζε την παραγωγή του. Αν αποφάσισε αρνητικά θα πήγαινε στο δικαστήριο. Ε, η Κομισιόν δεν αποφασίζει. Μα δεν επιτρέπεται αυτό. Αξιότιμη κυρία Μάγερ, ωραία αυτά που μας λέτε τα επιχειρήματα, αλλά δεν εξηγείτε γιατί. Πολλά τα βασίσατε σε μια αλλαγή, ανταλλαγή ελογραφία το 97, τα γνωρίζω. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, κάποιες παρεξηγήσεις που στα δικά μου μάτια έχουν ε, διασκεδαστεί. Ναι, ωραία. Ακόμα και αυτό να συνέβη. Γιατί από το 97 δεν κάνατε τίποτα μέχρι το 2007. Η οδηγία ορίζει ρητά το συντομότερο θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία τη ασφαλιστική ρήτρα. Τι θα πει για σα το συντομότερο, 10 χρόνια, αν δεν έχει αλλάξει τίποτα μέχρι σήμερα και ολοκληρωθεί. Και σα ερωτώ και με ενδιαφέρει, για σας ποια είναι η αρμόδια αρχή παρακαλώ. Στη Γερμανία είναι το κρατήδιο Σαξονία Άνχαλτ. Και εκεί γράφει ότι το 1996 υποβλήθηκαν όλα τα έγγραφα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και ε, αντιρρήσει. της Βαβαρίας μέχρι σήμερα δεν έχουν τακμηριωθεί και μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει τίποτα για τις συστάσεις αυτές, για την αρμόδια αρχή. Εσείς λέτε ότι δεν είναι αυτή η αρχή αρμόδια, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι. Γιατί θα θεωρώ όλα αυτά σημαντικά να σας εξηγήσω. 30 εκατομμύρια είναι στην Ευρώπη οι ασθηματικοί και εγώ έχω άσθημα από παιδί. 14 χρόνια. Αυτό που σας δείχνω με το δεξί μου χέρι είναι φάρμακο και αυτό που σας δείχνω το αριστερό είναι, λέγεται medical device. Είναι ε, μια συσκευή που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να πάρω το φάρμακό μου όπως οποιαδήποτε ένεση. Μπορεί να το, το βάλω σε αυτό ή στο άλλο. Αυτοί που κυριαρχούν την αγορά λένε ότι αυτά τα δύο μπορούν να πολλούνται μόνο μαζί. Παρόλο που το σπρέι είναι φάρμακο και μόλις τελειώσει το σπρέι πρέπει να πετάξω και τη συσκευή. Και υπάρχει ένας άλλος που το φτιάχνει πιο φτηνά, πιο αποτελεσματικά και λένε τα ταμεία ε, κερδίζουμε λεφτά, έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα, κανείς δεν έβαλε πρόβλημα και ένσταση και εσείς ε, δεν επιτρέπετε στον άνθρωπο αυτό να γνωρίζει τι γίνεται. Και θα πρέπει να λέμε κι εμείς ότι δεν μένουμε ικανοποιημένοι με απαντήσεις που δεν είναι ικανοποιητικές. Δεν θα επιτρέψουμε ένας κατασκευαστής να στερηθεί των δικαιωμάτων του. Βέρτμαν. Ευχαριστώ. Πολύ περίπλοκη η κατάσταση, το είπαν και οι προλήσαντες. Έχω ολόκληρο το εδώ γεμάτο έγγραφα και τα έγγραφα είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Το ένα λέει κλινικές μελέτες απαιτούνται και υποτίθεται ότι έχουν έρθει και οι κλινικές μελέτες. Μετά βλέπω ένα σημείωμα που λέει δεν είναι απαραίτητες οι κλινικές μελέτες και τελικά οι κλινικές μελέτες είναι απλή διπλωματική εργασία. Ε, τι γίνεται τότε, τι τρέχει, τι ισχύει. Και αν χρειάζονται κλινικές δοκιμές, ποιες δοκιμές ακριβώς χρειάζονται. Έχουν ε, κατατεθεί, αν όχι γιατί. Και αν ναι, γιατί δεν αναγνωρίζεται αυτό. Πολλά είναι τα ερωτηματικά για μένα. Έχουμε δύο προϊόντα ε, το εφέκτο και ένα άλλο που ταυτίζονται, δεν ταυτίζονται, οι ξυσαφίξεις, τι γίνεται τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Ναι, και εγώ το ελπίζω, απαντάει η ομιλήτρια στον κύριο Χέφνερ που δεν ακούμε γιατί είναι εκτός μικροφών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η νομική επιτροπή να ασχοληθεί σε λεπτομέρειες με το θέμα και να ψάξει και την κατάσταση και ό,τι αφορά τις υπόλοιπες λεπτομέρειες δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τους προαλήσαντες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Όκεν. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Υπάρχει κάτι τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, φρύση που υπόνουν. Εδώ ποιος δεν θέλει. Η φαρμακευτική βιομηχανία δεν θέλει. Γιατί θα χάσει πάρα πολλά χρήματα αν αυτό το προϊόν που χρησιμοποιεί λιγότερα φάρμακα εγκριθεί και περάσει στην αγορά. Θέλω να αποφεληθώ από την ευκαιρία αυτή για να σας πω ότι εδώ έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα της ανάγκης που υπάρχει να υπάρχει μητρό των διαφόρων λόμπι. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για την Πόρσε, έτσι, σε μια αναφορά η φαρμακευτική η βιομηχανία να ξέρετε ότι είναι τουλάχιστον εξίσου καλή λόμπιστ όπως και βιομηχανία. Να λοιπόν ένα ακόμα παράδειγμα που έχουμε και που δείχνει ποιοι κάνουν λόμπι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήταν μεγάλη απώλεια για την φαρμακευτική βιομηχανία αν ε, μπορούσε να πουληθεί αυτό το προϊόν. Βλέπω ότι δεν συμφωνεί η Κομισιόν, όμως ε, με συγχωρείτε. Ένα τέτοιο απλό σύστημα με τόσο απλή συσκευή θα έπρεπε να την εγκρίνετε. Τι είναι αυτά. Νομίζω ότι η, απόσταση της, ε, η απάντηση της Κομισιόν δημιουργήσε, έδωσε λαβή για πολλά σχόλια στα μέλη της Επιτροπής μας. Χρειάζεται λοιπόν μια σύνθεση. Παρακαλώ λοιπόν μία γραπτή απάντηση. Γραπτή της θέσης της Κομισιόν. Και θα ζητήσω από τον Επίτροπο Ντάλι να μας ε, διαβεβαιώσει λίγο, γιατί αυτό που ακούσαμε σήμερα είναι διαφορετικό αυτό που ακούσαμε τις προάλλες. απαιτούμε μια τελική απάντηση που θα επιτρέψει στον αναφέροντα πριν ε, ο αναφέρον χρειαστεί να προσφύγει σε άλλου είδους ένδικα μέσα. Μέχρι το Σεπτέμβριο πρέπει να έχουμε την απάντηση. Διαφορετικά ο Επίτροπος δεν θα είναι στο ύψος της υπόσχεσης που έδωσε. Ένα λεπτό έχει η Κομισιόν για να απαντήσει. Thank Σας ευχαριστώ. Ας πάμε πίσω στην αρχή. Η αρχική διαδικασία ήταν μια διαδικασία βάσει του άρθρου 8, διαδικασία ασφάλεια safeguard, που ξεκίνησε από το 97. Το εξέτασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άκουσε όμως ότι δεν υπήρχε πρόθεση από τον κατασκευαστή να προχωρήσει σε πωλήσει του προϊόντος. Θα ήταν καλό να είχε ρωτήσει η Επιτροπή, να είχε ζητήσει μάλλον από τη Γερμανία να αποσύρει την ρήτρα διασφάλισης. Δεν το έκανε γιατί δεν θεώρησε ότι χρειαζόταν. Εκείνη τη στιγμή πιστεύαμε ότι όλοι καταλάβαιναν. Όταν όμως επέστρεψε στην αγορά 10 χρόνια αργότερα το προϊόν, ενημερωθήκαμε από τον κύριο Κλάιν ότι υπήρχε άλλη απαγόρευση και κοιτάξαμε πολύ προσεκτικά την απαγόρευση αυτή και αποφασίσαμε ότι δεν ήταν διαδικασία του άρθρου 8, αλλά του άρθρου 18. Οπότε, από το 2005 και μετά, η... κοιτάξαμε τις διάφορες συνθήκες, προϋποθέσεις βάσει του άρθρου 18. Δεν ε, αφαιρέσαμε το δικαίωμα του κυρίου Κλάιν να προχωρήσει, το δείχνει αυτό εξάλλου και η διαδικασία στα γερμανικά δικαστήρια, τα οποία αποφάσισαν ότι το προϊόν έτσι όπως παρουσιάζεται σήμερα δεν ανταποκρίνεται στους όρους της φαρμακευτικής συσκευασίας. Τώρα αντίθετα με αυτό που είπατε εσείς, δεν υπάρχει κανόνες που λέει ότι δεν μπορεί να πουληθεί χωριστά το ένα κομμάτι από το άλλο, η συσκευή από το φάρμακο. Μπορεί κάλλιστα. Αρκεί να είναι ασφαλής αυτή η συσκευή και το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι αυτή η συσκευή δεν έχει αποδειχτεί ότι είναι ασφαλής. Ο κύριος Κλάιν λέει ότι είναι δύο φορές πιο αποτελεσματική γιατί το φάρμακο περνάει κατευθείαν στα πνευμόνια και ότι χρειάζεται η μισή δόση φαρμάκου για το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι το φάρμακο λειτουργεί διαφορετικά. Άρα πρέπει να αποδειχτεί ότι είναι ασφαλής αυτή η διαδικασία και ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνος να είναι η δόση λιγότερη ή να επικάθεται διαφορετικά στα πνευμόνια ή οτιδήποτε άλλο. Ας μην αρχίσουμε συζήτηση τώρα. Η διευκρίνηση αυτή δεν νομίζω ότι διασκεδάζει τις αμφιβολίες. Ε, παραμένουν ευφωλίες μας για τη συμπεριφορά της Κομισιόν επί του θέματος αυτού. Θα ζητήσουμε καταρχήν μία απάντηση από τον Επίτροπο Ντάλη και τα σχόλια ε, που μας έδωσε η, η εκπρόσωπος της Κομισιόν ζητάμε να μας δεθούν και γραπτά για να δώσουμε στον αναφέροντα να εξακολουθήσει αυτή ε, η καταντιμωρία διαδικασία. Το Σεπτέμβριο στους συντονιστές θα δούμε τι λύση θα επιλέξουμε. Κύριε Πρόεδρε, Νομίζω θα μπορούσατε να δώσετε στο τέλος το λόγο στον αναφέροντα, ίσως αυτό ξεκαθαρίσει λίγο το θέμα, αν του επιτρέψετε να μιλήσει. Αν. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ενδεχομένω και παρανόηση. Ένα λεπτό. Μην επαναλαμβάνω τα Ένα λεπτό μπορείτε να έχετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όντως, εδώ είναι η πλήρη συσύχηση που έχει προκαλέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και μου επιτρέπετε για το άρθρο 1, 8 και 18. Στις 22 Φεβρουαρίου του 2007 πατά ο Γενικός Γραμματέας επιστολή που λέει ότι είναι βάσει το άρθρο 8, εδάφιο 2 της αντίστοιχης οδηγίας. Τώρα το 18 πώς τους κατέβηκε, δεν καταλαβαίνω καθόλου. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρξει διαδικασία ασφαλιστική ρήτρα. Και σε ό,τι αφορά το βάρο τη απόδειξη, δεν μπορεί ο αναφερόμενο να αποδείξει ότι είναι ασφαλέ το προϊόν του. Το αντίθετο, αν το κράτο μέλο ε, θέλει να προσβάλλει το προϊόν και να προχωρήσει σε λήψη μέτρων, η οδηγία 9342 προβλέπει ότι το κράτος μέλος θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι επικίνδυνο. Δεν είναι δουλειά του κατασκευαστού να αποδείξει ότι είναι επικίνδυνο το προϊόν του. Κατά τα άλλα, έχει κάνει, έχει τις αποδείξεις και μόνο ότι τόσα εκατομμύρια χρήσεις έκτοτε έχουν γίνει από τους ε, ασθενείς και αυτό φυσικά αποδεικνύει ότι προφανώς είναι ακίνδυνο και ασφαλές. Και για τα πραγματικά περιστατικά, ποτέ κανείς δεν είπε ότι θα αποσύρει από την αγορά το προϊόν του και κανένας άλλος κατασκευαστής, έχουμε και τις αποδείξεις εδώ, ανέκαθεν κυκλοφόρησε ε, κυκλοφορούσε στο εμπόριο το προϊόν, δεν χρειάστηκε να αποσυρθεί ποτέ και για το διοικητικό δικαστήριο του Μονάχου για την επιστολή του κυρίου Τσούρεκ ε, ότι δεν βασίστηκε σε αυτή την επιστολή και αυτό είναι λάθος γιατί το λέει απόφαση ότι βασίστηκε. Αυτά ήθελα να ε, διευκρινίσω για λόγους αρχής. Ευχαριστώ. Είπαμε τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε αυτά τα κείμενα που ζητήσαμε και το Σεπτέμβριο θα αποφασίσουμε. Το θέμα παραμένει στην ημία συνδιάταξη. Περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η οδηγία Gold Stream στην Βαλτική. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ που πέρασε η συζήτηση αυτή σήμερα το απόγευμα, μια που δεν είχαμε χρόνο το πρωί. Είχαμε ψήφισμα του Κοινοβουλίου πριν από δύο χρόνια με συμπεράσματα τα οποία είχαν να κάνουν με την αξιολόγηση, ανεξάρτητη αξιολόγηση σχετικά με ένα μεγάλο σχέδιο πρωτόγνωρο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνέπειες είναι δυνατόν ε, να προβλεφθούν αν προηγουμένως δεν υπάρχει αυτή η ανεξάρτητη εξέταση. Πρόκειται για έναν αγωγό που φτιάχνεται. Ήδη ένα μέρος είναι έτοιμο. Το μήκος θα είναι συνολικά 220 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλο είναι αυτό το σχέδιο. Το Μάιο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στην Επιτροπή μας για το ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό σχέδιο και συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν αρμόδια για να κάνει την αξιολόγηση αυτή. Ε, βάσει της άποψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα έγγραφα που είχαμε στη διάθεσή μας από τη Φιλανδία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, Ινστιτούτα δηλαδή εκεί, ήταν πολύ καλά. Όμως, ο εργολάβος ο οποίος ζήτησε την αξιολόγηση αυτή, την ανάλυση αυτή, θεώρησε ότι δεν πρέπει να δεχτούμε αυτή την αξιολόγηση. Υπάρχει οδηγία του 1985 που επιβάλλει την υποχρέωση Αξιολόγηση αντικτύπου στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στο άρθρο 5. Αλλά μιλάει εκεί όχι μόνο για το δημόσιο τομέα, αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα. Το άρθρο 5 συγκεκριμένα αποτελεί ένα κατάλογο των στοιχείων της αξιολόγησης αυτής και μεταξύ άλλων μιλάει και για τις καταστροφικές συνέπειες που μπορούν να προκληθούν στο περιβάλλον εξαιτίας ε, τέτοιων ε, σχεδίων. Μιλάει μάλιστα και για το τι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση. Βάσει λοιπόν του άρθρου 5 της οδηγίας αυτής έχω κάποιες ερωτήσεις. Στο τεχνικό φάκελο που έχουμε της Nord Stream την ευθύνη σε περίπτωση οικολογικής καταστροφής στη Βαλτική θάλασσα δεν καθορίζεται συγκεκριμένα. Δεν λέει ποιος είναι υπεύθυνο, ποιος έχει την ευθύνη εναντίον ποιου θα πρέπει να στραφούμε. Έχουμε προηγούμενο πια στον κόλπο του Μεξικού. Στην περίπτωση της Βαλτικής θα μπορούσαμε να, βοηθήσουμε κλείνοντας τη ροή του φυσικού αερίου. Αν όμως υπάρξει έκρηξη στη Βαλτική, ποιος θα ήταν τότε υπεύθυνο για τις δραστηριότητες διάσωσης. Ποια από τις χώρες αυτές θα είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες αυτές διάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν διαθέτει μέσα για να δώσει εντολή για μια τέτοια μελέτη αντικτύπου. Υπάρχει όμως το πρόγραμμα Bonus με 50 εκατομμύρια ευρώ πρόβλεψη, πρόγραμμα για έρευνες στη Βαλτική θάλασσα. Ακριβώς για να αντιμετωπίζονται περιβαλλοντικές απειλές στη Βαλτική θάλασσα. Ε, περί αυτού πρόκειται λοιπόν εδώ. Πρόκειται για μια απειλή που έχουμε από την οποία κινδυνεύει το περιβάλλον. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί κάλλιστα μέσω του προγράμματος Bonus να χρηματοδοτήσει μια τέτοια αξιολόγηση αντικτύπου. Τελικά τα έχουμε αυτά τα χρήματα ή δεν τα έχουμε. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Στη σελίδα 30 του μη τεχνικού τμήματος της έκθεσης Nord Street λέει τα στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τις πιθανότητες διαρροής στον αγωγό δείχνει ότι η πιθανότητα αυτή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Άρα η απειλή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλή. Όμως, μιλάνε για κάποιες διαδικασίες που προβλέπονται στην περίπτωση που παρόλα αυτά υπάρξει κάποια διαρροή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ξέρει αυτή τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρακολουθήσει αυτές τις διαδικασίες. Είναι εν γνώση δεδομένου ότι ήδη υπάρχουν πολλά πράγματα στη Βαλτική θάλασσα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή λοιπόν η διαδικασία αντιμετώπισης κινδύνων από χημικές ουσίες που θα φτάνανε στη Βαλτική είναι γνώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τι κάνει με τη μη κύρωση από πλευράς της Ρωσίας μιας σύμβασης ΕΣΠΟ για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους διασυνοριακά. Στο τεχνικό τμήμα του εγγράφου ο υπογράφων αναφέρεται σε αυτή τη σύμβαση. Πώ είναι δυνατόν να κάνει μνήα τη σύμβαση αυτή εφόσον δεν την έχει συνυπογράψει. Ο Επίτροπο Δήμα, μάλιστα την παρουσία μα, είχε πει ότι θα υπήρξαν πιέσει από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ρωσία, ώστε η Ρωσία τελικά να επικυρώσει τη σύμβαση αυτή. Τι έγινε τελικά με αυτή την πίεση, υπήρξε ή είχε αποτέλεσμα, ξέρουμε τίποτα. Ένα άλλο ζήτημα τώρα αυτό το τεράστιο σχέδιο που κοστίζει και πάρα πολλά χρήματα προβλέπεται για 50 χρόνια. Μετά τι θα γίνει με την υποδομή αυτή. Ποιος θα είναι υπεύθυνο άπαξ και δεν χρησιμοποιείται πια για να ξεκάνει αυτήν την υποδομή και να τη διοχετεύσει. Θα είναι ασφαλής αυτή η διαδικασία. Η έκθεση Nord Stream δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Γι' αυτό θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου απαντήσει. Εξάλλου, πιστεύω ότι κάθε μας αμφιβολία που ήδη διατυπώθηκε πριν από δύο χρόνια, ισχύει ακόμα. Είναι μια μικρή θάλασσα, η Βαλτική θάλασσα. και ο κύκλος ε, ανταλλαγής νερού, δηλαδή από τη Βαλτική στον ωκεανό, παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Αν υπάρξει οικολογική καταστροφή σε μια τόσο μικρή λεκάνη όπως είναι αυτή της Βαλτικής, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για όλες τις χώρες και όχι μόνο για τις χώρες που συμμετέχουν στην κατασκευή του αγωγού. Η Λετωνία, η Λιθουανία, η Εστονία είναι και οι τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην το ξεχνάμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. τη Σάμπασης. Thank Ευχαριστώ και για την παρουσίαση του θέματος. Θα προσπαθήσω συντομία να συνοψίσω τη θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ψήφισμα αυτό και ε, στη συνέχεια θα ε, απαντήσω, θα προσπαθήσω τουλάχιστον να απαντήσω στα όσα ρώτησε η κυρία Βουλευτή. Αυτό το θέμα του North Stream είναι μια δραστηριότητα πάρα πολύ περίπλοκη και λόγω του μεγέθου και του δύο συνοριακού του χαρακτήρα. Αναφέρονται διάφορα σημεία στο ψήφισμα, ε, κυρίως περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αλλά έχουμε και άλλα για τον κίνδυνο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις εξωτερικές σχέσεις Ακούσαμε την περιβαλλοντική διπλωματία. Καταλαβαίνετε Κανονικά εδώ θα έπρεπε να είναι παρόντες ε, όλοι οι επίτροποι για να συζητήσουν αυτό το θέμα. Αλλά το βασικό ζήτημα για την Κομισιόν είναι ποιο ο θεσμικό τη ρόλο ω προ το σχέδιο αυτό και το έργο. Σύμφωνα με την οδηγία που αναφέρατε, 85337, που έχει σχέση με τη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου έργων ε, του δημοσίου αλλά και ιδιωτικών. Υπάρχει ένα πλαίσιο για τους διάφορους ε, εργολάβους και άλλους που κάνουν αυτά τα έργα με αντίκτυπο και είναι η ευθύνη του ε, εκτελούντος, είτε αυτό είναι ιδιώτης είτε είναι το δημόσιο. Υπάρχουν και εθνικές αρμόδιες αρχές που δίνουν ε, άδειες ε, ε, οικοδομής ή εκτέλεση ενός έργου. Και προηγουμένως ο βασικός στόχος της οδηγίας είναι να γίνει μια μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου και διαβουλεύσεις με το κοινό, με εθνικές αρχές και για διασυνοριακά έργα σαν αυτό εδώ, με τα κράτη-μέλη διαβουλεύσεις τα ενεχόμενα. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν σύμφωνα με την οδηγία αυτή που εφαρμόζεται και ψηφίστηκε και από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν είναι ούτε να δίνει την άδεια για την κατασκευή του έργου, ούτε να εκτιμά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ή να δει με ποιο τρόπο τα κράτη-μέλη μεταφέρουν και εφαρμόζουν την οδηγία. Αν διαβάσετε τα παραρτήματα, ε, είναι 100 ε, είδη έργων εμ εντατική κτηνοτροφία, αυτοκινητόδρομη, ε, αγωγή πετρελαίου φυσικού αερίου, ο δεν θέλησε να το δώσει αυτό στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι γιατί δεν μπορεί να τα ελέγξει, αλλά γιατί κυρίως είναι θέμα επικουρικότητας. Κατά πρώτο λόγο τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που είναι αρμόδια να ελέγξουν το έργο, τα, κράτη όπου γίνεται το έργο. Γι' αυτό απουσιάζει ε, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από εδώ δεν προβλέπεται ρόλος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να αναθεωρεί την οδηγία αυτή και τέλη Ιουνίου άρχισε μια δημόσια διαβούλευση με στόχο αναθεώρηση. Αν θέλει το Κοινοβούλιο λοιπόν να δώσει ένα ρόλο καινούριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις μελέτες σε όλα τα κράτη-μέλη, είστε προσκεκλημένοι ως μεμονωμένοι βουλευτές ή ως και Επιτροπή Αναφορών να μας δώσετε τις απόψεις σας. Αλλά το θέμα είναι η κείμενη νομοθεσία που πρέπει να εφαρμοστεί και τι μπορεί να κάνει βάσει αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρακτικά τίποτα. Στα κράτη-μέλη εναπόκειται να εγκρίνουν αυτό το project και αυτό συνέβη και στη βαρούσα περίπτωση. Η North Stream, η εταιρεία δηλαδή που έχει αναλάβει το έργο, προτίμασε μελέτες ε, ε, βάσει την εθνική νομοθεσία των κρατών από όπου θα περάσει ο αγωγός και έχει απευθυνθεί λοιπόν στις αρμόδιες αρχές των κρατών αυτών μελών συν τη Ρωσία και ετοίμασε και μια συνολική μελέτη εγκάρσια ξέρω εγώ, που προσπαθεί να αξιολογήσει όλο το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτή η συνολική μελέτη ε, έγινε μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να έχουμε συνολική θεώρηση του διασυνοριακού αυτού έργου. Λοιπόν, έχουμε μελέτες αντικτύπου και εθνικές και συνολικές. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές που έλαβαν και τις δύο μελέτες αυτές ε, ζήτησαν επιπλέον πληροφορίες από την εταιρεία, έγιναν και άλλες μελέτες και άλλες πληροφορίες και κυκλοφόρησαν για το κοινό όχι μόνο εκεί που περνούν ε, οι αγωγοί, αλλά και άλλες χώρες Βαλτικής και Πολωνία. Και βάσει αυτού, στα τέλη του 2009, αρχές του 2010, όλα τα κράτη-μέλη ενέκριναν την κατασκευή του έργου. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που δεν έχουμε μυστηρισμικό ρόλο, προσπαθήσαμε πρώτα απ' όλα να συμβουλεύσουμε και τα κράτη-μέλη και την εταιρεία για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το έργο, διασυνοριακό, δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί την πολιτική της ε, ισχύ, είτε με τεχνικές ε, συνεδριάσεις με ε, εμπειρογνώμονες από τα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά και με τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί υπάρχει και σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα διασυνοριακά έργα ή έργα με διασυνοριακό αντίκτυπο. Στα πλαίσια του ρόλου της λοιπόν και του περιορισμού του ρόλου προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει κάποια πίεση και να συμβουλεύσουμε τα κράτη-μέλη όποτε ετήθη το ζήτημα για το πώς να παίρνουν τις αποφάσεις. Και συνεχίζουμε γιατί υπάρχουν και άλλοι αγωγοί, ο ε, Ναμπούκο για παράδειγμα. Και αν θέλουν να ρωτάνε τα κράτη-μέλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα ερμηνευτεί η οδηγία αυτή του 85 για διασυνοριακά έργα, είμαστε εδώ για να ε, τους δίνουμε συμβουλές και μέχρι τα τέλη του έτους θα έχουμε και ένα κατευθυντήριο κείμενο, ένα οδηγό για να βοηθάει. Ε, συνοψίζω λοιπόν, παρόλο που δεν έχει θεσμικό ρόλο που να απορρέει από την οδηγία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και για να απαντήσω στις ερωτήσεις των βουλευτών για την ευθύνη. Υπάρχει η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη που βρίσκεται εδώ εφαρμογή, δηλαδή αν υπάρχει μεγάλη ζημία για το περιβάλλον, τότε μπαίνει αυτή η οδηγία και ο κατασκευαστής θα πρέπει να αποκαταστήσει τις ζημιές σε ό,τι αφορά τη Ρωσία και την σύμβαση ΕΣΠΟ. Ναι, την έχει υπογράψει αλλά δεν την έχει κυρώσει η Ρωσία τη σύμβαση αυτή. Ο Επίτροπος κύριος Δήμας και άλλοι επίτροπες, ε, επίτροποι πίεσαν τη Ρωσία και η λύση ήταν ότι δεσμεύτηκε de facto η Ρωσία να τηρήσει τις απαιτήσει της ΕΣΠΟ. Σε ό,τι αφορά τη Βαλτική και τους διάφορους κινδύνους εκεί είναι γεγονός ότι το περιβάλλον είναι πάρα πολύ εύθραυστο, έχουμε και στρατηγική για τη Βαλτική, αλλά επιπλέον και οδηγία για τη στρατηγική για θάλασσα που από το 2011 θα εφαρμοστεί και θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα και της Βαλτικής. Αν έχετε ερωτήσεις, είναι εδώ και άλλοι συνάδελφοι. Από άλλες γενικές διευθύνσεις θα σταματήσω εδώ όμως. Ε, Ευχαριστούμε. Αρχή συζήτηση. Παρακαλώ σαν δύο λεπτά ο καθένας. Βαλένσα. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις σας. Η Κομισιόν προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε το θέμα αυτό. Σας θυμίζω ότι το 2007 30.000 αναφορές ήρθαν στο Κοινοβούλιο για τον αγωγό αυτό κυρίως λόγω της ε, απειλής για το περιβάλλον, για τη Βαλτική. Ξέρουμε με μεγάλη πλειοψηφία 550 έναντι λίγων ψήφων εγκρίθηκε αυτό το σχέδιο στο Κοινοβούλιο και επισήμανε κινδύνους για την οικονομία, για το περιβάλλον, για τον καταναλωτή. Απαιτείται αξιολόγηση επιπτώσεων, ανεξάρτητη. Να την κάνει κάποιος που θα επιλεγεί από όλα τα κράτη της Βαλτικής. Δεν δόθηκε συνέχεια σε αυτό το ψήφισμα. Στην προηγούμενη συνεδρία ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μας είπε ότι υπάρχουν χιλιάδες σελίδων εμπειρογνωμοσύνης για το σχέδιο αυτό. Άρα η Κομισιόν δεν θα χρειαζόταν άλλα έγγραφα. Παίζουν με τη διαδικασία, παίζουν ένα παιχνίδι, γράφουν, κάνει η Κομισιόν εδώ. η Κομισιόν ως εκτελεστική εξουσία θα έπρεπε να υλοποιεί τις συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Να υποβάλει την υλοποίηση του προγράμματος αυτού στη Διεθνή Συνθήκη για το δίκαιο της θαλάσσης και άλλους συναφείς περιβαλλοντικούς κανόνες. Πρόσβαση στα πολωνικά λιμάνια στη Βαλτική και ρωτώ. Είπατε εκπρόσωπος Λέιδη Άστον πότε θα έρθει να συζητήσει με το Ευρωκοινοβούλιο για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος να ακούσουμε τη θέση της. Τονίζω μια φορά ακόμη ότι μια πολύ περίεργη κατάσταση μπορεί να είναι κανείς υπέρ ή κατά του προγράμματος αυτού. Εδώ όμω πρόκειται για τη μη τήρηση των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, λεπόμενος ομιλητής. Συμφωνώ και εγώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Εδώ και δύο χρόνια το Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισε ένα ψήφισμα με συγκεκριμένα στοιχεία και συστάσεις προς την Κομισιόν. Ένα μεγάλο μέρος από αυτά δεν υλοποιήθηκε. Όπως το Κοινοβούλιο είπε ότι να μην γίνουν οι επενδύσεις στην κλίμακα που προβλεπότανε αν δεν έχουμε μελέτη επίπτωση στο περιβάλλον και ζήτησε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο να την κάνουν αυτή την ανάλυση του αγωγού αερίου τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν προϋποθέσεις για, την, για γνωμοδότηση εκ μέρους Κομισιόν όπως προβλέπει το άρθρο 6.4 της Οδηγίας 9243. Η Κομισιόν έπρεπε κάτω το Κοινοβούλιο να κάνει μια αξιόπιστη τέτοια αξιολόγηση μελέτη, να δει τα βιομηχανικά απόβλητα και άλλα προϊόντα που ρηπαίνουν την Βαλτική και τι άλλα προβλήματα θα δημιουργούσε το πρόγραμμα Nord Stream. Έπειτα θα πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικέ διαδρομέ για τον αγωγό αερίου για λόγους περιβάλλοντος και οικονομικούς. δυστυχώ, ούτε αυτές οι συστάσεις εισακούστηκαν. Σα θυμίζω το Ευρωκοινοβούλιο δεν ήταν το μόνο που πήρε αυτή τη θέση και η Επιτροπή Αναφορών και η Επιτροπή Εξωτερικών και οι Ήτρε ασχολήθηκαν. Είναι δυνατόν ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου να τα αντιμετωπίζει με τέτοια περιφρόνηση και ασέβεια η Κομισιόν διότι είναι ανεξάρτητη και αξιόπιστη η μελέτη επιπτώσεων που την πλήρωσε ο επενδυτής α, εδώ υπάρχει σύγκρουση φερόντων, σοφός. Εμείς ζητήσαμε τα πράγματα να γίνουν με αντικειμενικό τρόπο. Έπειτα δεν μελετήθηκαν οι χερσαίες διαδρομές που θα συνδέουν την Ρωσία με τις χώρες μέλη. Αυτό θα στήχιζε λιγότερο. Και ρωτώ την Κομισιόν. Αυτές τέτοιου είδου σχέσεις θέλει η Κομισιόν με το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Αναφορών, αλλά της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Οι συζητήσει αυτές λοιπόν με ενδιαφέρουν πολύ, γιατί πριν από τρία χρόνια εκπροσωπούσα μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι οποίες απευθύνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με την αναφορά αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε ότι έχει πολιτική βούληση και προχώρησε με τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε πριν από δύο χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως σιώπησε και η σιωπή αυτή είναι πολύ απογοητευτική. Για το σχέδιο αυτό λοιπόν, όταν ρωτάμε για τον Nord Stream την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε πάντα την ίδια απάντηση. Ότι είναι ένα καθαρά εμπορικό σχέδιο δύο χωρών και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, το σχέδιο αυτό μπήκε στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Έχει αυτό το καθεστώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπώς, έτσι εμπλέκεται σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που ζητάει η αναφορά είναι μία ανεξάρτητη αξιολόγηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, να δούμε μήπως υπάρξουν ε, αντισταθμίσματα για την ε, ζημιά στο περιβάλλον ή μήπως υπάρχουν ε, άλλες εναλλακτικοί οδοί. Τίποτα δεν έγινε. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που υπόθηκε και πριν, ότι θέλουμε μια αξιολόγηση αντικτύπου, ανεξάρτητη εντελώς. Και τώρα θα έρθω λίγο στο τι γίνεται για το περιβάλλον. Το φθινόπωρο του 2009 στη Βαλτική θάλασσα έγιναν έρευνες βάσει του 169 πόνου που έδειξαν ότι τα τοξικά επίπεδα στη θάλασσα παντού στον κόλπο της Φιλανδίας και στο νότιο τμήμα της Βαλτικής είναι 10 φορές παραπάνω από τα κανονικά επίπεδα. 8.000 για παράδειγμα σε ε, ρέγγα. Καταλαβαίνετε ότι το ζήτημα τίθεται, γιατί δεν συγκρίνουμε τις έρευνες 2000, 2001, 2004, τα στοιχεία αυτά είναι τα ίδια. Ενώ τώρα, το 2009, τα τοξικά επίπεδα αυξάνουν φοβερά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, μπορεί να βρει έναν τρόπο να ελέγξει το σχέδιο. Γιατί όταν ρωτάμε την Όρθιν ποιος ευθύνεται για τη ζημιά, στην αρχή έλεγαν ότι έχουν αρκετά χρήματα και τώρα λένε ότι υπεύθυνοι είναι οι χώρες που δίνουν τις άδειε. Οπότε τελικά είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το λεγόμενο ιδιωτικό σχέδιο. Ο κ. Βορτινάρο. Κυρία Πρόεδρε, πρώτον, ευθύ εξ αρχής θα σας πω ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένο από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα το πρωί είδαμε ότι έχει διπλέα, δύο μέτρα και δύο σταθμά η Επιτροπή. Σήμερα το πρωί μας είπε ναι, μα γίνανε λάθη, γίνανε σφάλματα, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Στην περίπτωση της πολυεθνικής της Πόρσε και τα εμπορικά του συμφέροντα. Τώρα μας λένε ότι υπάρχει νομικό κενό και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει και να κάνει αυτήν την περιβαλλοντική αξιολόγηση αντικτύπου. Μα κύριε Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βρίσκεστε εδώ σήμερα, μετά την καταστροφή του κόλπου του Μεξικού, όταν η British Petroleum αναγκάστηκε 20 δισεκατομμύρια δολάρια έβαλε για να αποζημιώσει. Και ξέρετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση σήμερα για την BP. Ε, λοιπόν, εσείς Πώς μπορείτε να μας καθησυχάσετε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε μια αντίστοιχη κατάσταση. Έχουμε τους οικονομικούς πόρους να καλύψουμε κινδύνους και καταστροφές ενδεχομένως εάν πτωχεύσει ο επενδυτή στο μέλλον. Πείτε μου, πώς. Πώς μπορεί ο επενδυτή να καλύψει το κόστος. Τι θα μας πείτε, συγγνώμη δεν έχω απάντηση, εν πλήρη ηρεμία. Δεύτερον, πριν από δύο μέρες ο Επίτροπος πατρότη μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία θα αλλάξει ακριβώς παίρνοντας μαθήματα από την καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού. Και εσείς έρχεται σήμερα και μας λέτε εντάξει δεν έχουμε αρμοδιότητα, είναι εμπορικό το σχέδιο. Και με κάθε ηρεμία έρχεται και μας λέτε, φιλικά βέβαια, ότι η Ρωσία είπε πως θα τηρήσει τη σύμβαση. Ξέρετε τίποτα για την ε, στρατηγική για τις επαφές Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Δεν νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να πιέσει τη Ρωσία για να επικυρώσει την ε, σύμβαση ΕΣΠΟ. Εδώ τι έχετε να απαντήσετε σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών. Πάλι θα πείτε συγγνώμη. Είναι απαράδεκτες αυτές οι απαντήσεις. Εν κατακλείδη. Τελικά, εάν μια τέτοια μαρτυρία ερχόταν στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε οι αντιπρόσωποι εκεί, να ξέρετε, δεν θα δεχόταν κάτι τέτοιο. Δεν θα δεχόταν με τίποτα αυτά που λέει σήμερα σε μας εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παίζει μαζί μας. Είναι απαράδεκτο αυτό το παιχνίδι. Να το περάσετε στους επιτρόπους αυτό το μήνυμα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσετε να παίζετε αυτό το παιχνίδι. Κοροϊδεύετε εγώ δεν είμαι κατά του σχεδίου. Και στην ε, Μαύρη Θάλασσα θα έχουμε Nord Stream, Ναμπούκο, ίσως και τα δύο. Αλλά πείτε μου, τι θα κάνουμε με την Ρωσία όταν έχουμε μόνο τη Ρουμανία και τη Βολγαρία εκεί. Δύο μικρές χώρες με τόσο λίγη επιρροή. Πώς. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει τις ευρωπαϊκές αξίες εκεί στον εύξενο πόλο. Πώς πάλι θα είναι μια έτσι γλυκιά και ήρεμη απάντηση. Για μας όμως είναι απαραδεκτή. Ευχαριστούμε κύριε Μποσινάρο. Η συνάδελφος Γκέρνιερ για τα συμπεράσματα. Παρακαλώ σύντομο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως βλέπετε δεν μας ικανοποιεί η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν θα σταματήσουμε να ρωτάμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ερώτησή μου που πιστεύω ότι είναι η πιο σημαντική και περιμένω να με καθησυχάσετε. Ποιος θα είναι υπεύθυνο εφόσον χρειαστεί μια διάσωση. Είναι πέντε χώρες που επενδύουν στο σχέδιο αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι το φυσικό αέριο κανονικά είναι η διοκτησία της Ρωσίας όσο δεν έχει φτάσει στη Γερμανία. Οπότε ας υποθέσουμε ότι προκαλείται από τον αγωγό ε, μία καταστροφή, το αέριο ανήκει στη Ρωσία, σας ρωτάω ποιος θα ευθύνεται για τις αποζημιώσεις και για τη διάσωση. Είναι μια ερώτηση που χρειάζεται απάντηση. Την περιμένουμε αυτή την απάντηση βάσει του άρθρου 5 που αναφέρεται στους τρόπους διάσωσης στον ιδιωτικό τομέα. Θέλουμε αυτή την απάντηση. Ε, λόγω του ότι δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι, παραμένει το θέμα ανοιχτό και αναβάλουμε για αποφάσεις που θα πάρουμε το Σεπτέμβριο. Θέλει κάποιος να μιλήσει. Ο συνάδελφος. 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα επίσημα να ζητήσω από την Κομισιόν μετά την αυστηρή κριτική που ασκήσαμε της θυμίζω το ψήφισμά μας η Κομισιόν να εφαρμόσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου ένα δεύτερο ψήφισμα θα ήταν χρήσιμο και δικαιολογημένο νομίζω με βάση τη δερμία κριτική που ασκήθηκε στο, στην Κομισιόν, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να προσφύγουμε σε ένα δεύτερο ψήφισμα. Πρόεδρος. Πρέπει να δοθεί συνέχεια που μου έστειλε ο κύριο Λεβίνσκι και που έστειλε στον πρόεδρο Μπούζεκ και ζητάει να δοθεί συνέχεια στην απόφαση του Κοινοβουλίου για λόγους αξιοπρέπειας και του, του θεσμού και των αξιών που αντιπροσωπεύουμε θα αποφασίσουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας τι θα κάνουμε στους συντονιστές. Το επόμενο. Έκθεση για την επισκέψη εξεταστικής αποστολής στην Καμπανία. Έχουμε τον ε, ε, εκπρόσωπο από την Ιταλία που ήρθε και που κάθεται δίπλα μου. Έχουμε τους αναφέροντες. Επειδή έχουμε πάρα πολλούς παρόντες, παρακαλώ κατά κεφαλή ένα λεπτό, αν μιλήσετε όλοι, ή τέσσερα λεπτά, αν μιλήσει ένας για όλους. Πέντε λεπτά μας είπαν ότι μπορούμε να μιλήσουμε. Είμαστε δύο. Δύο είμαστε. Τρία λεπτά λέτε. Έχουμε ένα πρόβλημα χρόνου. Έχουμε ήδη καθυστερήσει κατά μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά. αν θέλουμε να πάρουμε μέρος και εκπρόσωποι των Κομισιών, ο εκπρόσωπος της Ιταλίας και να τους ακούσουμε όλους, θα πρέπει ο καθένας να είναι λακωνικός. Πρακτικό είναι το θέμα. Αν είστε τέσσερι, δύο λεπτά ο καθένας, μαξιμο. Ο κύριος Εσπόζη το πρώτος. Επειδή ο έμφας Μέρκες, η συνάδελφη Γιάννη και η κυρία Όκεν θέλουν να μιλήσουν. Θα κάνουν αυτή την εισαγωγή. Θα τα πω δανέζικα. Μάλιστα. Να τα πείτε. Λοιπόν, έχουμε μια έκθεση στα αγγλικά και στα ιταλικά αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν διάβασα τις δύο αυτές εκδοχές, είδα το δανεικό κείμενο. Και αυτά που λέει είναι πάρα πολύ θετικά και ευνοϊκά απέναντι στις αρχές. Ε, δεν είχαμε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα όταν ήμασταν επί τόπου. Θέλω πρώτα να συγκρίνω τις ε, μεταφράσεις πριν σας πω την τελική μου θέση. Έχουμε δει το, πρόγραμμα, το πρόβλημα από όλες τις πτυχές, από όλες τις πλευρές του το είδαμε σφαιρικά, είδαμε ποια είναι τα παράπονα και οι καταγγελίες και ας πω το εξή, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι η κρίση αυτή δεν έχει λυθεί καθόλου μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα σαφές σημάδι ότι θα γίνουν σεβαστά τα όσα ορίζει η οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων, ότι θα μειωθούν τα απόβλητα και θα αυξηθεί η ανακύκλωση, όλος αυτός ο σχεδιασμός που θα έπρεπε να έχει γίνει δεν έχει γίνει. Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι για να λυθεί το πρόβλημα της αποκομιδής των ε, αποβλήτων στην καμπανία χρησιμοποιούσαν χωματερές. Τελεία. Ε, περιβαλλοντική μελέτη και τα λοιπά τα αποφύγανε γιατί ήταν σε ανάγκη και είπα αφού είναι κατεπήγον δεν χρειάζεται κανένα κριτήριο και ε, καμία προδιαγραφή. Δεν προλαβαίνουμε. Ναι, εντάξει, αλλά εμείς πού να καταλάβουμε τι γίνεται όταν πάμε εκεί ως αντιπροσωπεία. Δεν μπορούμε να δηλώσουμε αν είναι ικανοποιητική η κατάσταση. Είπαμε ότι σε μερικά σημεία που γινόταν αποτέφρωση, δεν υπήρχε διαχωρισμός των σκουπιδιών που πήγαινε στον αποτεφρωτήρα. Είδαμε μέχρι και βαρέλια με χημικές ουσίες που απαγορεύεται να ε, καίγονται ως απόβλητα. Οπότε η κατάσταση χρειάζεται καλύτερο σχεδιασμό και μάλιστα μακροπρόθεσμο για να ε, υποστηρίξουμε και περαιτέρω χρηματοδότηση. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά δεν είδαμε πολλά βιομηχανικά απόβλητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμαρτύρεται, αλλά στην έκθεση είδαμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διακίνηση ε, ε, βιομηχανικών αποβλήτων, όχι μόνο από τη Βόρεια Ιταλία, αλλά και από αλλού. Στη συνέχεια δεν πήγαμε στις παράνομες χωματερές. Υπάρχει επιθυμία για ε, περισσότερη αποτέφρωση των αποβλήτων, αλλά και αυτό είναι προβληματικό από μόνο του, ως επιθυμία. Δηλαδή όλα τα απόβλητα δεν προσφέρονται για αποτέφρωση. Ας ελπίσουμε λοιπόν να μας δώσουν πιο ικανοποιητικές απαντήσεις οι Ιταλικές αρχές. Εμείς δεν πρόκειται, λοιπόν, αν δεν δούμε καλό σχεδιασμό, να συμφωνήσουμε να δοθούν και νέα κονδύλια. Ένα σχεδιασμός που να εμπνέει εμπιστοσύνη. Έχουν χαθεί πολλά λεφτά στην καμπανία και κοινοτικά χρήματα για την διαχείριση των αποβλήτων με πάρα πολύ ε, πενιχρά αποτελέσματα. Σήμερα δεν ήμουν προετοιμασμένη να τα πω όλα αυτά. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω μπει σε όλες τις λεπτομέρειες. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι άξιζε τον κόπο η επίσκεψη εκεί. Κάναμε καλές επιθεωρήσεις ε, μαζί με τους συναδέλφους μας εκεί και τους Ιταλούς και την κυρία Μασόνη βεβαίως και ελπίζω στη διαδικασία αυτή και στη σημερινή συζήτηση με τον αναφερόμενο και τους άλλους ε, παρόντες. Ελπίζω λέγω τελικά μετά τη συζήτηση αυτή το Σεπτέμβριο να το ξανασυζητήσουμε. Θα έχουμε και εκπρόσωπο της υπηρεσίας περιβάλλοντος και αυτοί έχουν εμπειρία για το πώς λιώνεται τέτοιου είδους προβλήματα γιατί η Ιταλία δεν είναι μόνη της. Λοιπόν, ελπίζω το Σεπτέμβριο να έχουμε καλή προσέγγιση και αποτέλεσμα. Δεν, είναι καλό να, δεν αρκεί να έχει μια καλή έκθεση και μια καλή παρουσίαση. Λύσει πρέπει να δίδονται. Όχι μόνο στην Καμπανία, γενικότερα στην Ιταλία. Και ο Πίτερ Γιάρη ήταν εκεί και αν νομίζει ότι κάτι ξέχασα παρακαλώ να συμπληρώσει. Έχει και άλλα σχόλια, φαντάζομαι, Πίτερ Γιάρ. Αν έχει, ε, παρακαλώ να τα κάνει. Grazie, ο συνάδελφος Γιάν θα παρέμβει μετά, αφού μιλήσουν οι αναφέροντες. Προηγουμένως όμως ο εκπρόσωπο της Κομισιόν, Ζουζέπε Μαγκανάρα. Ευχαριστώ. Ως εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης για το Περιβάλλον, να σας ε, πω δύο λόγια που βρισκόμαστε σήμερα με τη διαδικασία παράβασης σχετικά με τα απόβλητα, στην διαχείριση των αποβλήτων στην καμπανία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, πήρε απόφαση στις 4 Μαρτίου και είπε ότι στην καμπανία υπάρχει πρόβλημα ε, ανεπαρκούς διαρθρωτικής ανεπάρκειας όσον αφορά τη διαχείριση. Στις 23 Μαρτίου η Κομισιόν έστειλε επίσημη επιστολή στις Ιταλικές Αρχές και ζητάμε πληροφόρηση για το τι μέτρα προβλέπει να υιοθετήσει ή υιοθέτησε η η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου. Η επίσημη απάντηση των Ιταλικών αρχών μας ήρθε τον περασμένο μήνα. Την αναλύουμε, την αξιολογούμε χωρίς να θέλω να προδικάσω τα αποτέλεσματα αυτής της ε, ενέργειας, είναι σαφές για μας ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στα εξή δύο. Πρώτο θα ζητήσουμε από τις Ιταλικές αρχές και από τις αρχές της καμπανίας να αρχίσουν να εφαρμόζουν ένα περιφερειακό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων που θα πρέπει να εγκριθεί και από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Κομισιόν και θα ζητήσουμε από τις Ιταλικές Αρχές να μας δώσουν και ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την υλοποίηση υποδομής που χρειάζεται να είναι επαρκές το δίκτυο αποβλήτων. πότε προβλέπεται η κατασκευή και η λειτουργία των μονάδων αυτών. Επίσης θα επιμείνουμε στο θέμα του κομπάλ. Πρέπει να γίνει προσαρμογή των μονάδων στην Ιταλία έτσι ώστε να υπάρχει και τα νέα απόβλητα που παράγονται καθημερινά να μπορούν να τα διαχειριστούν αλλά ταυτόχρονα να λυθεί μια για πάντα και το πρόβλημα των ιστορικών αποβλήτων, όσε ορί που έχουν δημιουργηθεί. Χρονοδιάγραμμα λοιπόν δράσης. όπου με αξιόπιστο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσει, αντιμετωπίσει και το πρόβλημα των κομπάλ. Ευχαριστώ. ο κύριος Ρώμα από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή. Εγώ θα μπορούσα να σας αναφέρω τα κονδύλια. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο προγράμματα. Το ένα από το 2000-2006 συνολικό ποσό υπέρ του περιφερειακού συστήματος αποβλήτων 170 εκατομμύρια 50% από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάλυσης, ε, Ανάπτυξης. Στις 27 Ιουνίου του 2007, 29 Ιουνίου του 2007, ε, στάθηκε αιτιολογημένη γνώμη και μπλοκαρίστηκαν τα κονδύλια. Περίπου 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα παραμένουν μπλοκαρισμένα τα κονδύλια αυτά. Οι Ιταλικές αρχές έκαναν προσφυγή στο πρωτοδικείο η απόφαση του πρωτοβάθμιου αυτού δικαστηρίου προβλέπεται να βγει στο τέλος του 2010. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελικά νούμερα για το 2000-2006 θα οριστικοποιηθούν στην τελική έκθεση που θα πρέπει να στείλει η περιφέρεια της Καμπανίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 30 Σεπτεμβρίου 2010. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να τα γλιτώσει τα χρήματα αυτά η περιφέρεια διότι είναι δυνατόν να περάσουν τα χρήματα σε κάποιο άλλο τμήμα και να απορροφηθούν. Καθαρά λοιπόν όπως προβλέπουν όπως βλέπει η τελική έκθεση, ο απολογισμό, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα υπάρξουν ε, απώλεια, καθαρό απώλεια κονδυλίων κοινωτικών χρημάτων. Ωστόσο παραμένουν μπλοκαρισμένα. Η δεύτερη περίοδος, 2006-2013. Και εδώ υπάρχουν κονδύλια για τη διαχείριση των αποβλήτων 270 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Από αυτά, για αυτά τα χρήματα μάλλον, υπάρχει μια ρήτρα που προβλέπεται στο πρόγραμμα Τρεις όροι τίθενται. Ο πρώτος, τον είπε ο συνάδελφος από το περιβάλλον, Πρώτος όρος είναι εκβανών, είναι ότι η καμπανία θα στείλει ένα περιφερειακό πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων επίσημα και η Κομισιόν Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα το μελετήσει και θα το εγκρίνει. Δεύτερος όρος είναι οι έκτακτες μονάδες και οι έκτακτες διαδικασίες να σταματήσουν. Τυπικά το Υφυπουργείο για το αρμόδιο σταμάτησε να λειτουργεί. Αλλά επειδή η έκθεση του, όπως λέει η έκθεση, η έκθεσή σας, για φέτος μπορεί ακόμα ε, ε, ένα επιπλέον έργο να εκτελεστεί από άλλες υπηρεσίες έκτακτα. Από τη στιγμή που θα μας υποβληθούν αποδείξεις για πληρωμή, αν πληρείται ο πρώτος όρος, θα ζητήσουμε οι περιφερειακές αρχές να μας επιβεβαιώσουν, να πιστοποιήσουν ότι η διαδικασία, ιδιαίτερα για την εξολόγηση επίπτωση περιβάλλοντος και τη διαδικασία των διαγωνισμών, ότι όλες συμφωνούν με την κοινωτική οδηγία. Υπάρχει και ένας τρίτος όρος. Από τη στιγμή που οι αρχές στην καμπανία αιτιολογήσουν τη δαπάνη, θα ζητήσουμε από τη διαχειριστική αρχή να επιβεβαιώσει οι δαπάνες αυτές για τις οποίες ζήτησαν, ζητήθηκε αποζημίωση, συμφωνούν με τους στόχους του προγράμματος. Από τη στιγμή που οι περιφερειακές αρχές θα μας προτείνουν επιστροφή χρημάτων, σίγουρα θα συμφωνούν με τους στόχους του προγράμματος. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. Οι αναφέροντε. Ο κύριος στο δύο λεπτά. Είναι σημαντική η προσοχή του Κοινοβουλίου μέσω της Επιτροπής σας επειδή υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για το σοβαρό πρόβλημα, έκτακτη ανάγκη των σκοπιδιών στην Καμπανία. Η προσπάθεια να τα κρύψουμε και να τα κουκουλώσουμε τους τελευταίους μήνους θα αποτύχει, όπως έχουν διαπιστώσει ο τύπος και στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Τίποτα δεν γίνεται για να μειωθεί η ποσότητα των σκοπιδιών που πάει στις χωματερές και στους αποτεφρωτές. Μέχρι στιγμής μόνο λόγια λόγια και προθέσεις. Στην αποστολή σας που ήρθατε τον Απρίλιο στην Καπανία για να σας καθησυχάσουν για να περιφερώσετε τα κοινωτικά κονδύλια που έχουν παγώσει μετά την απόφαση του Ευρωκαθιστηρίου που καταδίκασε την Ιταλία που δεν ενέκρινε για την Καμπανία επαναλαμβάνω τα κονδύλια μπλοκάριστηκαν λόγω της απόφασης του Ευρωδικαστηρίου και η αντιπροσωπεία σας δεν είδε αυτό το δίκτυο το οποίο έχετε ζητήσει να συσταθεί ακόμα στην Ιταλία, στην Καπανία ούτε και αλλού στην Ιταλία δεν υπάρχει. Πολλές φορές που ήρθαμε και μιλήσαμε εδώ και υλικό που δόθηκε στην αντιπροσωπεία στην επίσκεψή σας. Μιλάμε μόνο για τους αποτεφρωτήρες απορριμμάτων. Όσο πιο πολλά καίγονται, τόσο πιο πολλή ενέργεια, τόσο πιο πολλά χρήματα αφαιρούνται από τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Το να πληρώνουν εξακολουθούν να είναι οι πολίτες από την τσέπη τους για τα σκοπίδια. το 7% του κόστος για τον πολίτη του ηλεκτρικής ενέργειας πάει στους αποτεφρωτήρες. Για όλα αυτά, το κόστος δηλαδή που πληρώνουν οι πολίτες, η έκθεση της αντιπροσωπείας για όλα αυτά δεν λέει τίποτα. Στο πρόγραμμα 2010-2013 μόνο λόγια και κατευθύνσεις αναφέρονται. στο Σαλέρνο, στην Νάπολη, στη Σάντα Μαλέρνο και θα γίνει κι άλλος ένας από τη Και ο πρόεδρος της επαρχίας του Μπενεβέντο ζητάει να γίνει άλλη μία μονάδα. Όλα αυτά είναι παράλογα. Αυτό παραβιάζει και την οδηγία 2006 αλλά και την τελευταία οδηγία του 2008 της Ένωσης που προβλέπει την αρχή της ιεράρχησης στην ε, καταστροφή των απορριμμάτων. Η πρόταση του να αποτεφρώνονται τα σκουπίδια δεν λύνει το πρόβλημα. Η πλειοψηφία από τις τελευταίες εκλογές δεν έφεραν ένα νέο στοιχείο όπως προσπάθησαν να σας κάνουν να πιστέψετε. Τα τελευταία χρόνια όλα τα μέτρα που εγκρίθηκαν έγιναν με συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών. Αυτός που κυβερνάει σήμερα ή χθε την περιφέρεια είναι ο ίδιος που κυβερνάει σήμερα ή χθε την Ιταλία. Για τη χωματερία του Βερτσίνου τίποτα δεν έγινε. Και όποιος δίνει μάχη σήμερα να, να κλείσει η χωματερία αυτή δεν έκανε τίποτα άλλο για να κλείσει κάποια άλλη. Πριν από λίγες μέρες, άλλοι με περίπτωση πολίτες που φωτογραφίζανε τη χωματρή του σκηνή τους σταματήσανε. Δεν έχουμε διάλογο, δεν έχουμε αλλαγή. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν είναι αλήθεια. Μάλλον οι πολίτες κατάλαβαν τη φιλοσοφία της αποτέφρωσης. επέκριναν αυτή την επιλογή, ζητάνε ανακύκλωση των απορριμμάτων και όμως κανένας δεν τους ακούει. Ένα σωρό ψέματα. Άρα δεν πρέπει να παρατηθούμε. Ο κύριος λόγος της κρίσης της καμπανία περνάει μέσα από το πάση θυσία να γίνουν οι νέοι αποτεφρωτές. Άλλο είναι ο ιδιοκτήτης, άλλος είναι ο διαχειριστής της μονάδας αυτής. Και υπάρχουν εγγύησεις τραπεζών που χρηματοδότησαν την επένδυση αυτή. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί η αντιπροσωπεία σας. Ενώ αναγνωρίζει τα απορίσματα ότι έγινε η μονάδα αυτή χωρίς οι πολίτες να έχουν τρόπο να πάρουν πληροφορίες για το κατά πόσον τηρούνται οι προδιαγραφές αξιολόγηση επίπτωσης για το περιβάλλον δεν λέει τίποτε για τη δραστηριότητα αυτή απόσβεσης του έργου με βάση τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν, παραμένουν σοβαρές, σοβαροί ενδιασμοί σχετικά και με το προϊόν που μπαίνει στο ποτεφυτήρι και με το προϊόν που βγαίνει και την τοξική στάχτη. Το περιβάλλον ήδη βρίσκεται σε κίνδυνο όπως επίσης και η υγεία του πολίτη. Και βάζουμε και τα πρακτικά μιας απαγόρευσης βοσκής, ελεύθερης βοσκής ζώων στην περιοχή πριν αρχίσουν να λειτουργούν οι απορρεφωτήρες. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο της αρχής της καμπανίας του Ιουνίου του 2010 όπου αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία εξυγίανση του εδάφους έτσι ώστε να σταματήσει η απαγόρευση τη ελεύθερη βοσκή Και ορίζεται εκ νέου η μη δυνατότητα απαγόρευσης ελεύθερη βοσκής λόγω διοξίνη από την άρπαξη των παρατηρητήριων πάνω στοιχεία για τις 28 Μαρτίου του 2009 Τέλος Δεκεμβρίου ο πρόεδρος λέει ότι πρέπει να τελειώνετε γιατί δεν έχετε χρόνο. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει υπέρβεση των αξιών στη σκόνη στην περιοχή. Στη βιομηχανική περιοχή της Ατσέρα ε, ο νόμος προβλέπει 35 μέρες το χρόνο το πολύ υπέρβαση. 112 μέρες είχαμε υπέρβαση. πώς είναι δυνατόν ένα παρατηρητήριο στο οποίο συμμετέχει ο διαχειριστής της μονάδας είναι δυνατόν να δώσει εγγύηση στους πολίτες. Αυτό ορίζει τους ελεγκτές. Η επιδημιολογική μελέτη, τι γίνεται, πού είναι. Είναι δυνατόν να περιοριστεί ο δήμαρχος της ΑΣΕΡΑ να μην μπορεί να στείλει άτομα στο παρατηρητήριο. Πρόεδρε, σας ζητάμε ένα ελάχιστο σεβασμό. Δέκα λεπτά μιλάτε. Εμείς δεν συμφωνούμε. Θα επαγρυπνούμε. Κυρία Πρόεδρε, εμείς ερχόμαστε από την Ιταλία με δικά μας έξοδα Νομίζω, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ το Κοινοβούλιο, νομίζω είναι δίκαιο να μας δώσετε τη δυνατότητα να εκφραστούμε με ένα ελάχιστο πληρότητας αυτό που ζούμε στο πετσί μας εδώ και χρόνια. Δεν είναι δίκαιο να μην μας δώσετε αυτή την ευκαιρία. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίε πολιτικοί, πρόεδρος. Ευχαριστώ. Το τελευταίο σχόλιο ήταν ε, δεν υπήρχε λόγος να γίνει. Είμαστε στη διάθεση όλων των αναφερόντων εμείς. Εμείς δεν μπορούμε όμως και να ξεπεράσουμε μια μερίσια διάταξη η οποία ορίζεται από την αρχή του χρόνου και μοιράζεται με θέματα κατά μήνα. Γιατί υπάρχουν και άλλοι πολίτε, όπω εσεί που έχετε από τι άλλε 27 χώρε τη Ένωση, που έχουν και αυτοί το δικαίωμα να ακουστεί η φωνή του. Σα είπα, μία ώρα για το θέμα αυτό είναι επαρκής. Αν εσείς μόνο σας πάρετε 12 λεπτά, δεν θα υπάρχει χρόνος για όλους. Θα ήταν πιο χρήσιμο να ήσασταν λακωνικός προς το συμφέρον σας των πολιτών, να προσθέσετε τα νέα στοιχεία που υπάρχουν για να μπορούμε να έχουμε πιο πλήρης απαντήσεις. Δεν είναι χρήσιμο να έρχεται εδώ να κάνετε μια διακήρυξη. Την κριτική την ακούω. Προσπαθώ να κάνω τη δικά μου όσο πιο καλά γίνεται. Για να Μαρκίδη Ταρανιέρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Πρόεδρο και όλη την Επιτροπή για που μου δίνετε το λόγο και τους ε, βουλευτές που ήρθανε τον Απρίλιο στην καμπανία για να δούνε με τα μάτια τους την πραγματικότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εγώ θα μιλήσω απλά. Και το, το, το, το επιλέγω αυτό για να είμαι σαφής. Εμείς λέμε ο πιο κουφός είναι αυτός που δεν θέλει να ακούσει. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Εκεί που ζούμε και από εκεί που ερχόμαστε η αναφορά για τη χωματερή του Τερτσίνιο έχει 3.500 υπογραφές των κατοίκων του Τερτσίνιο, Μποσκορεάλε, Μποσκοτρεκάσε και Τρεκάσε. Τέσσερις κοινότητες. Οι πολίτες πάντα ήταν κατά της χωματερής αυτής μέχρι το 2007 όταν έγινε μια πρώτη πρόταση μέσα στο Εθνικό Πάρκο του Βεζουβίου ενός χώρος που η ίδια η Ένωση αναγνώρισε κοινοτική σημασία και ειδική ζώνη προστασίας με την Οδηγία 9243 και την απόφαση της Κομισιόν του 2006. 613. Η χωματερή δηλαδή έγινε σε ένα χώρο ο οποίο έπρεπε να είναι προστατευμένο και με βάση την Ιταλική νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή. Αντίθετα, βλέπουμε να ρίχνουν αδιαφοροποίητα, όχι ξεδιαλεγμένα δηλαδή απορρίμματα πριν πάνε στη χωματερή, αλλά με διευρύνεται η χωματερή. υπάρχουν εγκάρσεις ενισχύσεις με τσιμέντο της χωματερής για να μπορεί να πέσει περισσότερο υλικό. Ευχαριστώ όλη την αντιπροσωπεία που ήρθε τον Απρίλιο και την πρόεδρο Ματσόνη βέβαια. και την κυρία Όκεν και άλλον έναν ευρωβουλευτή γιατί αυτά που είπατε με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι. Εμείς θέλουμε ο πλήρης κύκλος των απορριμμάτων να έχει σωστή διαχείριση με βάση ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ιταλικές προδιαγραφές. Γιατί εμείς οι πολίτες του Τερσίνιου και των γειτονικών κοινοτήτων και της Καμπανίας δεν είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους. Είμαστε πολίτες ίσοι όσο και όλοι οι άλλοι και αυτή τη μεταχείριση θέλουμε όχι να ζούμε συνέχεια πολίτες έκτακτης ανάγκης. Ένα πράγμα ακόμη. Επειδή έχουμε τον κύριο Ρωμάνο εδώ, δεν ρωτώ. Η εφημερίδα Ιλματίνο της Νάπολη το πρωί δημοσίευσε μία συνέντευξη του πρόεδρου της καμπανίας Καλντόρο, όπου ο Καλδόρο ζητάει να ξανακηρυχθεί η έκτακτη ανάγκη για τα απορρίμματα στην Καμπανία. Ζητώ εξηγήσει για τη συνέντευξη αυτή του πρόεδρου της Καμπανίας. Αν όντω αυτά τα είπε, αυτό δεν συμφωνεί με αυτό που είπε στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε στον κύριο Ρωμάνο την δυνατότητα να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να περιορίσω την απάντησή μου στο χρόνο που μου έχει δοθεί. Εγώ δεν θα μιλήσω, λέει ένας άλλος κύριος. Ε, Καλά, μετά μπορεί. Ε, έχουμε δυσκολία με το χρόνο. Στις 5 θα πρέπει να έχουμε τελειώσει αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να ακούσουμε το Σύμβουλο... Ναι. Αν θέλετε, ε, να ακούσετε και τα αντιπιχειρήματα. Θέλετε να ακούσετε το Σύμβουλο. Έχουμε τα υπέρ, τα κατά, να μην ακούσουμε την άλλη πλευρά. Δεν διάβασα σήμερα το πρωί την εφημερίδα της Νάπολης Δεν ξέρω αν ζήτησε και πάλι να κηρυχθεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, δεν συμφωνώ. Δεν είναι καθόλου η δική μας στρατηγική αυτή, ούτε αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε στη διαχείριση ενός ολοκληρωμένου κύκλου ε, διαχείρισης αποβλήτων. Ε, νομίζω ότι ουσιαστικά υπήρχε το εξής ε, σοβαρό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που θέτει ο νόμος 26 ε, του 2010 που ήρθε να τροποποιήσει το νόμο 126 του 2009. Αν ε, δούμε την κείμενη νομοθεσία και την τηρήσουμε, η διαχείριση των αποβλήτων από την 1η Ιανουαρίου 2010 περνάει στα χέρια των περιφερειών. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε. Πώς θα γίνει δυνατό κάτι τέτοιο μέσα σε πέντε μήνες να έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να αρχίσει αυτό να ισχύει από την 1η πρώτη 2010. Γι' αυτό ε, προτάθηκε παράταση ενός έτους για να ε, μπορέσουν οι περιφέρειες να ανταποκριθούν. Οι δήμοι και οι κοινότητες θεωρούν ότι αυτό το μοντέλο διαχείρισης με ένα και μόνο διαχειριστή δεν αντιστοιχεί στις απαιτήσεις των πολιτών και επίσης δεν αντιστοιχεί στην αποτελεσματικότητα που χρειάζεται για μια τέτοια υπηρεσία. Δεν είναι το ίδιο η ενιαία διαχείριση, γιατί η διαχείριση θα πρέπει βεβαίως να ολοκληρωθεί, να ενοποιηθεί. Τώρα έχουμε νομοθεσία για τις επικράτες, για τις περιφέρειες και πέντε περιφερειακές εταιρείες που κατέθεσαν ένα βιομηχανικό ε, πρόβλημα, πρόγραμμα συγγνώμη, για τη διαχείριση των αποβλήτων. Για την αποτέφρωση και μόνο μιλώ αυτή τη στιγμή. Η αποκομιδή των αποβλήτων, οι χωματερές παρεμένουν στα χέρια της τοπικής αυτοδίκησης για ένα χρόνο ακόμα. Για ποιο λόγο? Είναι προφανές ότι αυτό που ζητούν οι αναφέροντες και επίσης εξήγησε ο κύριος Μαγκανάρου και ο κύριος Ρώμα δείχνει σαφώς ότι οι τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να έχουμε ολοκληρωμένη διαχείριση είναι πρώτον ένα περιφερειακό πρόγραμμα ολοκληρωμένου κύκλου διαχείρισης αποβλήτων ε, Βαρό στη συνέχεια ένα περιφερειακό ε, πρόγραμμα, μάλλον για τα στερεά απόβλητα, το άλλο για τα ειδικά απόβλητα και ε, ε, για τα λίματα ας πούμε και για τα καυσαέρια. Γιατί και εκεί θα πρέπει στην Ιταλία να μεταφέρουμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Όλα αυτά λοιπόν συμπεριλαμβάνουν όλα τα ζητήματα και όχι μόνο τη διαχείριση των αποβλήτων. Πώς να βελτιώσουμε το νερό, πώς να βελτιώσουμε το έδαφος, αν δεν ξέρουμε τι ουσίες υπάρχουν στο νερό και το έδαφος. και από πλευράς προγραμματισμού. Τους δύο τελευταίους μήνες επιταχύναμε σημαντικά και έχουμε ένα πρόγραμμα περιφερειακής διαχείρισης ειδικών αποβλήτων. Ένας ερευνητικός οργανισμός της Καμπανίας, ανεξάρτητος, ε, συνεργάστηκε για την εκπόνηση αυτού του περιφερειακού προγράμματος. Είμαστε τώρα στη φάση της ενημέρωσης αυτού του προγράμματος και η νομοθεσία προβλέπει να εγκριθεί από τις περιφερειακές αρχές. Θα το κάνουμε αυτό την άλλη εβδομάδα. Είναι μακρά η διαδικασία βεβαίως, γιατί μετά θα πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο στο σύνολό του να εγκρίνει το πρόγραμμα. Πάντως, έχουμε κάνει ένα του δρόμου. Και για τα ειδικά απόβλητα, το σχέδιο που είναι σημαντικό, αντιπροσωπεύει 10.000 με 12.000 τόνους ημερησίως. Καταλαβαίνετε. Αλλά αν δεν υπάρχει ειδική διαχείριση για τα ειδικά απόβλητα, κινδυνεύουμε να μπούμε στην κατάσταση που διαπιστώσατε κι εσείς όταν ήρθατε στην καμπανία, ότι τα ειδικά απόβλητα είναι αναμεμειγμένα με τα στερεά αστικά απόβλητα, που είναι τα οικιακά απορρίμματα, βασικά τα σκουπίδια τα κανονικά. Αν δεν έχουμε ε, διαχωρισμό των αποβλήτων, στην πηγή είναι όλα χίδιν και τάκτος ερημένα. Θα πρέπει να διαχωρίζονται από τα οικιακά απόβλητα, τα ειδικά αυτά απόβλητα. Αυτά είχα να σας πω και τελειώνω εδώ. Συμφωνώ όταν μιλάτε για ολοκληρωμένη συνολική διαχείριση των αποβλήτων. Δεν ξέρω εάν είμαστε ήδη σε θέση να ανιστρέψουμε την τάση αυτή. Μπορώ όμως να σας πω ότι προσπαθούμε να το κάνουμε εγώ προσωπικά στα πλαίσια των ε, δικών μου αρμοδιτήτων. Δυστυχώς και αναλαμβάνω τις ευθύνε μου. Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Ο κύκλος διαχείρισης έτσι όπως έχει μας υποχρεώνει να συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε ε, τους δύο αποτεφρωτήρες της ε, Νάπολης και του Σαλέρνο. Η Επιτροπή Αναφορών άκουσε το έτοιμά σας, αλλά η χωματερή ε, του Καβαντιτέλο δεν πρόκειται να ανοίξει, γιατί γνωρίζουμε ότι μας χρειάζονται 3 εκατομμύρια κυβικά χώρος. Γιατί τόσα είναι τα απόβλητα που δεν μπορούμε να διαθέσουμε. Τρία εκατομμύρια κυβικά. Ορίστε, τι μας κληροδότησε η πολιτική προστασία. Έκλεισαν δύο αυτές χωματερές. Εντάξει, θα πρέπει να σεβαστούμε το νόμο 90 που πλέον ονομάζεται 123, είναι νόμος του Ιταλικού κράτους και προβλέπει δύο χωματερές χιτά στο Σαλέρνο και τη ε, Νάπολη, στην ε, επαρχία της Νάπολης στο Ταρσίνιο που ήδη έχει δύο χωματερές. Αρνούμαστε λοιπόν να ανοίξει και τρίτη χωματερή εκεί. Είμαστε σε ε, μόνιμη επαφή με τις τοπικές αρχές και για τη μασερία επίσης έχουν εκεί χωματερή και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο διαχωρισμός των αποβλήτων είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο για να γίνει συνείδηση, για να αλλάξουν οι συνήθειες, η νοοτροπία του κόσμου. Έχουμε απέναντί μας δημάρχους, τοπικούς άρχοντες που ακόμα δεν έχουν καταλάβει την ουσιαστική ε, σημασία του διαχωρισμού των αποβλήτων. Που εκεί είναι η ρίζα του προβλήματος. Σήμερα πάρα πολλοί πολίτες δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να διαχωρίζουν τα σκουπίδια τους. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να αρχίσουν προγράμματα διαχωρισμού των αποβλήτων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η κούρσα της επιδότησης, της χρηματοδότησης, όχι. Κονδύλια προβλέπονται για να γίνουν αυτά τα έργα, αλλά και πάλι κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε εμπλοκή διότι αυτή η υλικοτεχνική υποδομή έχει καθυστερήσει. Όλα αυτά τα προγράμματα κινδυνεύουν, επαναλαμβάνω, να οδηγηθούν σε εμπλοκή γιατί έχουν σταματήσει οι πληρωμές. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα έργα πλέον. Η περιφέρεια της καμπανίας δεν είναι σε θέση να προκαταβάλει τους απαραίτητους πόρους και το θέμα δεν είναι ότι θέλουμε οπωσδήποτε να βρούμε χρηματοδότηση και διψάμε για την επιδότηση. Όχι. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να βεβαιωθούμε ότι θα συνεχιστούν τα έργα. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια του στρατηγικού στόχου μέσω πρόθεσμα και με το, το Βάλε Λαμασερία και το Τερσίνιο, τις δύο χωματερές μπορούμε να πούμε ότι έχουμε βραχυπρόθεσμα πρόβλημα, διότι παράγονται κάθε μέρα 7.200 τόνοι ε, αποβλήτων. Αυτό είναι το πρόβλημα, οξύ, την ημέρα 7.200 τόνοι. Και μετά θα δούμε τη συνολικότερη στατηγική για να κτίσουμε το χαμένο χρόνο. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Συμπροματικά προς τη συνάδελφο Άουκεν για την αποστολή στην καμπανία. Τρία είναι τα θέματα που διαπερνούσαν πάντα τη συζήτηση έτσι ως ένας μύθος της Αριάδνης. Το πρώτο ήταν η αλήψη του διαλόγου. Και είναι καλό πάντα να συζητάμε και στους δύσκολους καιρούς. Και τα μέσα ενημέρωσης είναι εκεί για να καταδεικνύουν τα προβλήματα, να, τα εντοπίζουν, αλλά όχι να τα λύνουν. Για να τα λύνουν ο διάλογος. Το δεύτερο είναι η έλλειψη της διαφάνειας. Συχνά είχαμε το εξή φαινόμενο. Έλεγε η μία πλευρά το α, η πλευρά β. Η μία πλευρά έλεγε ότι υπερβαίνουν τα όρια και η άλλη πλευρά όχι, τι κατώτατε τιμέ. Τότε λέει ο σιωπηρό παρατηρητή αυτό που χρειάζεται είναι διαφάνεια. Να έχουμε δημόσια στοιχεία, ε, διαφανή και λύνεται το θέμα επιστημονικά και τελειώνει. Δεν υπάρχει λόγος συζήτηση. Αυτό είναι μεγαλύτερη διαφάνεια. Και το τρίτο, το είπε ο προλαλής σας. Εκτός από την βραχυπρόθεσμη στρατηγική, γιατί χρειάζεται μια διαχείριση τώρα των αποβλήτων ε, για το οξύ πρόβλημα, μετά θα πρέπει να υπάρξει και μια βιώσιμη στρατηγική πιο μακροπρόθεσμη. Και αξίζει τον κόπο. Υπάρχουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διατίθενται τα κονδύλια αυτά. Είναι δεδομένο αυτό. Βέβαια αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε ένα συνολικό σχεδιασμό και να καταργηθούν να κλείσουν οι παράνομες χωματερές. Ευχαριστώ και την Πρόεδρο και τους Ιταλούς συναδέλφους για τη διοργάνωση αυτής της αποστολής καταφέραμε να πάμε παντού όπου ήταν σημαντική η παρουσία της διερευνητικής των πραγμάτων αποστολής. Υποσχόμαστε στους ε, αναφερομένους ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουμε τις προθυρίες μας. Πάντα θα πιέζουμε και θα ρωτάμε γιατί είναι πολύ σημαντική να υπάρχει μια υφόρος διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων και να λυθεί οριστικά αυτό το θέμα. Είμαστε σε μια πρώτη φάση των εργασιών που χάρη στην πρόεδρο Ματσόνη και στους συναδέλφους τους μη Ιταλούς που ήρθαν με μας στην καμπανία στην Ιταλία. Ξεκίνησε μια θετική σχέση με τις επιτροπές, με τους αναφέροντες, επιτροπές πολιτών Πρέπει να κλείσουμε θετικά αυτό που συζητάμε σήμερα. να γίνει ένας έλεγχος του πώς θα έχει κατάσταση μετά από μερικούς μήνες. Και λέω για τον ε, κύριο Ρωμάνο, πρέπει να υπάρχει συνέπεια και μία ανακολουθία σε όλα τα θεσμικά επίπεδα. Στου επόμενου μήνε θα είναι πιο δύσκολο να κάνουμε αναφορά στο παρελθόν και θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο αναφορά στο παρόν. Τι θέλουμε να κάνουμε το ε, Ιταλικό Κοινοβούλιο και η Γερουσία μέσω ενός ε, βουλευτή από το Σαλέρνο ενέκρινε μία τροπολογία, δύο τροπολογίες μάλιστα, τώρα που συζητάμε, που ε, δημιουργούν δυσκολία στη δική μας δουλειά. Λέω δική μας γιατί εγώ είμαι συμμέτοχος σε αυτή τη δουλειά που γίνεται. Δηλαδή ενέκρινε μία, μία τροπολογία που λέει ο, η μονάδα στην Ατσέρα 350 εκατομμύρια κτίσει με κονδύλια όχι από, από τα περιφερειακά κονδύλια ΦΑΣ. Και το λέω σε εσά εκπρόσωπο της Ιταλίας γιατί από τα 350 εκατομμύρια 300 πηγαίνουν στο περιβάλλον και ειδικά για τα απορρίμματα. Υπάρχει κίνδυνος, ένα μεγάλο τμήμα από τα χρήματα αυτά να πάνε στην θερμομονάδα. Κανονικά θα πρέπει να πληρώσει η κυβέρνηση αυτή. Χρειάζεται λοιπόν κοινή δουλειά για να πείσουμε και τον βουλευτή αυτό από το Σαλέρο να αποσύρει αυτή την τροπολογία. Τουλάχιστον ο τύπος αυτό λέει ότι έκανε και να μην κάνουμε τέτοιου είδου δώρα σε αυτή την περίοδο. Δεύτερον, αν δούμε τι γίνεται με το σύμφωνο σταθερότητα, μπαίνει ένα επιπλέον στοιχείο. Πέρα από τα 5 ή 10 εκατομμύρια που έχουν μπλοκαριστεί και θα δοθούν ενδεχομένω κάποια στιγμή κλπ. Έχουμε το κριτήριο ότι μπλοκάρονται όλες οι υποχρεώσεις πληρωμών το τελευταίων 12 μήνων, όχι από τα κανονικά κονδύλια, αλλά από τα κοινωτικά κονδύλια, ουσιαστικά θα μπλοκαριστούν χρήματα που δεν έχουν σχέση με αυτά που συζητάμε. Εξυγίανση, υγιής κλπ. Εσείς πήρατε το αεροπλάνο, ήρθατε εδώ και ενώ σου ταξιδεύατε είχαμε αυτές τις δύο τροπολογίες στην Ιταλική Γερουσία. Μην παίζουμε τον παπά, όπως λέμε, με τα τρία χαρτιά που είναι ο παπάς. Αν πραγματικά θέλουμε να βρούμε διέξοδο και μην ξαναρθούμε στις ε, Βρυξέλλες εδώ να λέμε ιστορίες και παραμύθια όπως κάνουμε τα τελευταία δέκα χρόνια. Ιωβένε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Την ιστορία τη τα μεταγενέστερη. Είχαμε μια τραγική διαχείριση των απορριμμάτων. Ο κύριος Ρωμάνο ήρθε την περασμένη φορά εδώ και μας είπε ότι ναι, δεσμεύομαι, αλλά η καλή προαίρεση πολλές φορές δεν αρκεί. Δύο λόγια για την έκθεση της Επιτροπής μας. το λένε ακούσαν και οι αναφέροντες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η έκθεση αυτή δεν φωτογραφίζει αυτό που είδε η αντιπροσωπεία στην καμπανία. Ναι, πρέπει να δούμε τα απορρίμματα στον, σε ένα πλήρη κύκλο διαχείρισης. Συχνά τα ξεχνάμε αυτά στην καμπανία. Και όπως είπε μια κυρία από τους αναφέροντες που ανάφερε πριν. Εγώ θέλω να είμαι Ευρωπαίος πολίτης. Θέλω κάτι που δικαιούται ο φυσιολογικός πολίτης. Το ίδιο λέω και εγώ. Οι νέες περιφερειακές αρχές δεν θα μπορούν για πολύ καιρό να κυβερνάνε, να ελέγχουν μάλλον το φαινόμενο αυτό μετα... κοιτώντας προς το παρελθόν. Να κοιτάξουμε προς το μέλλον. Κύριε Ρωμάνο, ξέρω ότι εσείς είστε άνθρωπος σοβαρός που δεσμεύεστε και για μια φορά ακόμη στην Επιτροπή μας σας εύχομαι το έργο που θα επιτελέσετε να είναι επιτυχές. Πρόεδρος, ο κύριος Ρωμάνο σε τρία λεπτά φεύγει. Θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό μάλλον το Σεπτέμβριο πάλι. Η κυρία Άουκερ. Συμφωνώ να συνεχίσουμε το Σεπτέμβριο. Πάντως θέλω να ξεκαθαριστούν δύο πράγματα. Πρέπει να πούμε ότι η καλύτερη επικοινωνία δεν κοστίζει τίποτα, μόνο καλή βούληση. Και όπως είπε και ο Πιτυγιάσε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έλλειψη επικοινωνίας και μια πολύ κακή αντιμετώπιση των ανθρώπων που υποφέρουν από αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι κάτι που εύκολα μπορεί να διορθωθεί. Προς την Επιτροπή θέλω να πω ότι από την Επιτροπή δεν ακούω καθαρά κατά πόσο είναι διατεθειμένη να πάνω στα σοβαρά όλη την ιεραρχία για τα απόβλητα. Γιατί όταν ακούτε τους ε, και κυρίως από αυτά που είδαμε μπορεί να υπάρχουν ένα σωρό πουλιά στη σκεπή. Αλλά όταν φτάνουμε στην πραγματικότητα είναι θέμα στρατηγικής για την αποτέφρωση και για τους χώρους υγειονομικής ταφής. Και όταν συναντηθήκαμε με το Διευθυντή στη μονάδα αποτέφρωσης, είπε ότι όλα μπορούμε να τα κάψουμε. Και από τη Δανία, που ξέρω, έχουμε πολλέ τέτοιε μονάδε αποτέφρωση, δεν μπορεί να κάψει οτιδήποτε. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικό με το τι βάζει ακόμα και σε ένα μικρό αποτεφρωτή. Αν δεν γίνει αυτή η διάκριση για να ξέρουμε τι βάζουμε, κάνουμε πολύ κακό στο περιβάλλον και στον κόσμο. Και τα είδαμε αυτά στην πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω ότι ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο προσεκτική γι' αυτό. Και έχω και μια πρόταση. Δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε κάποια συγκριτική μελέτη για το τι γίνεται σε άλλες πόλεις. Πώς αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα άλλες πόλεις. Έτσι μπορούμε να έχουμε μια ιδέα του τι πρέπει να γίνει. Θα είμαστε πιο συγκροτημένοι με αυτόν τον τρόπο νομίζω. Η συνάδελφος Ντεμπράν ήθελε να παρέμβει, ζήτησε το λόγο. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τους συναδέρφους για την δουλειά τους. Είναι μια πολύ δυνατή έκθεση που σοκάρει. Σοκάρει να ακούει κανείς όπου υπάρχει μια κατάσταση όπου υπάρχει έλεγχος από το στρατό, ότι η αστυνομία δεν ε, μπορεί να δράσει. Τα είδα αυτά αντιπροσωπεία μας. Ο κόσμος θέλει να κοιτάει προς το μέλλον, όμως κρατείται μυστικός ο ρόλος του στρατού που θα παραταθεί για άλλον ένα χρόνο. Η έκθεση επίσης μιλάει για κατευθυντήριες γραμμές που υιοθέτησε η καμπανία για τη διοχέτευση των αποβλήτων αλλά αυτά είναι ίδια όπως και με την προηγούμενη δίκηση. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, αφού μας είπαν ότι θα υπάρξουν χρήματα για τη νέα μονάδα, λαμβάνεται υπόψη αυτό. Με το νέο πλαίσιο απαιτείται μέχρι αύριο 16 Ιουλίου να έχουμε τα νέα στοιχεία. Γιατί όλες τις χώρες... Εγώ δεν άκουσα τίποτα σήμερα που να λέει ότι αυτά που συζητάμε εδώ ευθυγραμμίζονται στις απαιτήσει που υπάρχουν για αύριο. Εδώ ακούμε ότι στοιχεία κλειδί της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας έχουν παραβιαστεί. Και δεν άκουσα τίποτα στη σημερινή συζήτηση μια ξεκάθαρη πρόταση για το πώς θα βγούμε από αυτό το διέξοδο. Δεν μπορούμε λοιπόν να είμαστε σε μια κατάσταση που λέει ότι αφού τόσο χάλια ήταν η κατάσταση μέχρι τώρα, ε, αν τώρα είναι λίγο καλύτερα, δηλαδή αντί να είναι πλήρως καταστροφική κατάσταση, είναι απλώς καταστροφική, ε, εντάξει, είναι καλό. Ε, όχι, δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να πούμε έντονα ότι πρέπει να υπάρξει έλεγχος προσεκτικά και ότι δεν δεχόμαστε μια τέτοια κατάσταση σαν και αυτή που σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεχτεί, να δώσει χρήματα και πάλι όταν υπάρχει τόσο ξεκάθαρη παραβίαση. Στη σελίδα 10 λέει κάτω-κάτω ότι και για τον αποτεφρωτή και για τον χώρο υγειονομικής αρχής δεν ζητήθηκε αξιολόγηση λόγω του κατεπήγοντος. Μπορεί, απαιτείται όμως η αξιολόγηση αυτή βάσει της οδηγίας 85337 και θέλω λοιπόν να ξέρω τι γίνεται, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αν εγώ πάω και εδώ στην αυλή του σπιτιού μου να φτιάξω έναν αποτεφρωτή, μπορώ. Δεν μπορώ. Εδώ λοιπόν πρόκειται για παράβαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Τι γίνεται λοιπόν τώρα για να αντιμετωπιστεί αυτή η παράβαση. Αυτές είναι απαντήσεις που χρειάζονται απάντηση και πρέπει να συνεχίσουμε το Σεπτέμβριο με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Βοποτζάνη, στον κύριο μάλλον Βοποτζάνη, συντάκτη για να συνοψίσει. Ο κύριος Ρωμάν έφυγε. Δεν είναι σωστό αυτό που είπε, ότι για να λυθεί το πρόβλημα των σκουπιδιών στην Καπανία πρέπει να γίνουν δύο αποτεφρωτήρες σήμερα για να δίνουν δύο προτιφτήρες χρειάζονται ε, πέντε χρόνια ενώ η διαφοροποιημένη αποκομιδή θα γίνει. Ας αρχίσουμε σήμερα με την διαφοροποιημένα απορρίμματα με μονάδες κομπόστ, με διαχείριση εμψυχρό για να γίνουν μονάδες εμψυχρό που υποκαθιστούν τους ε, χρειάζονται ελάχιστα εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν ήδη μονάδες στην καμπανία, τα περίφημα CDR, που κάνουν αυτές τις μεγάλες μπάλες οι οποίες πηγαίνουν στον απορτεφρωτήρα που είναι, έχουν γεμίσει τον τόπο μπροστά στα σπίτια του κόσμου, δίπλα στα χωράφια που καλλιεργούμε και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν όλες αυτές οι μπάλε. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο κατασκευής χωματερών και αποτεφρωτήρων, ας ζητήσουμε από την Ευρώπη τα χρήματα αυτά να αποδεσμευτούν μεν, αλλά για κατασκευή ενός σωστού κύκλου απορριμμάτων που εμείς οι επιτροπές το λέμε εδώ και έξι χρόνια. Αν στην περιοχή αυτή, στην Καμπανία, κάποιος μας είχε ακούσει τους τρελούς που υποστηρίζουν, που προστατεύουν τη γη τους τις επιτροπές μας, ίσως τώρα να μην ήμασταν σε αυτές τις συνθήκες που είμαστε. Ο κύριος Ρωμένα ειλικρινά μπορεί να είναι ο πιο καλός άνθρωπος στον κόσμο, αλλά δεν μπορεί να μας λέει ο κύριος Ρωμάνο ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, την ευθύνη έξι εκατομμυρίων ατόμων στην καμπανία πρέπει να είναι όχι στα χέρια ενός ανθρώπου. Ζητάμε την εφαρμογή της οδηγίας ΑΟΣ που λέει ότι μονά, όσον αφορά την διάθεση των σκουπιδιών, των απορριμμάτων, από κοινού οι αποφάσεις θα πρέπει να παίρνονται με τους πολίτες, με τις κοινότητες. Μέχρι σήμερα οι πολίτες δεν αποφάσισαν τίποτα. Εγώ, καλό και πάλι, την Κομισιόν, την πρόεδρο Μαντσόνη που μου κάνει την τεράστια ευχαρίστηση να έρθει στις 11 η ώρα το βράδυ, να έρθει στο Καγιάνο. Εμείς είμαστε στην Επιτροπή του Καγιάνο. Προσπαθήστε να κοιμηθείτε σε όποιο σπίτι, σε όποιον είναι σπίτι του Καγιάνο, 250.000 άνθρωποι που τη νύχτα δεν καταφέρουν να κοιμηθούν γιατί υπάρχει μια τεράστια βρώμα τεράστια βρώμα και δυσοδεία. Είχαμε και το Φερντινάντο που αυτός ήταν ο αναφέρον. Ελπίζω το Σεπτέμβριο να μπορέσει να μιλήσει και αυτός. Στο μεταξύ η Ευρώπη να στείλει ένα μήνυμα. Ο κύριος Ρωμάνο αν πραγματικά θέλει να υλοποιήσει τις προθέσεις του, ας καταφέρει να κάνει ένα περιφερειακό νόμο με βάση το οποίο οι βιομηχανικές αυτές μπάλε οι οποίες έρχονται προς αποτέφρωση να μειωθούν. Η, η, η Ευρώπη μιλάει για ανακύκλωση, νέα χρήση, μονάδες ανακύκλωσης και στο τέλος τέλος αν υπάρχει χωματερή και αποτεφρωτήρας στην καμπανία έχουμε το αντίστροφο χωματερή και από τεφροτήρες μόνο και από κάτω τίποτε. Και στη χωματερή του Κογιάνου και σε άλλες χωματερές έγιναν πάνω σε παράνομες χωματερές που τις έκανε η Καμόρα. 10.000 τόνοι αμίαντο από τα έλεγξε ο στρατός. 10.000 αμίαντος από κάτω. Και εκεί απάνω κάνανε μια χωματερή από την κυβέρνηση σε ένα δάσος που είναι πατρογονική κληρονομιά της Καμπανίας με τα πιο πολλά νοσοκομεία στο Νότο. Έξι νοσοκομεία σε απόσταση μέγιστο 2,5 χιλιόμετρα από τη χωματερή του Καγιάννα. 2,5 χιλιόμετρα συνοψίζω, γιατί ποτέ δεν μπορέσαμε να συνοηθούμε. Ποια είναι τα κριτήρια. Τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω. Συγγνώμη που μιλάω λίγο με έξαψη, αλλά πραγματικά έχουμε μεγάλη οργή με τις τελευταίες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Ρωμάνου, τι μας λέει. Θα αυξήσουμε τις χωματερές στην Νάπολη, Καγιάνο και Τερτσίνιο, γύρω από το Βεζούβιο. Όλοι οι ευρωβουλευτέ, αν πάρουν μια χάρη της Νάπολης βλέπετε, βλέπετε γιατί μιλάμε. Πιο γνωστές εικόνες της Ιταλίας Από τη μια μεριά θα μεγαλώσει η χωματερή στο Βεζούβιο, που είναι πατρική κληρονομιά της UNESCO, της UNESCO. Όλοι ξέρουμε πόσο ωραία είναι ο Βεζούβιος και η Νάπολη. Και από την άλλη θα μεγαλώσουν και άλλες χωματερές γύρω από τα νοσοκομεία, γύρω από τα σπίτια μας. Και θέλουν να κάνουν και από φροντήρες. Συγγνώμη, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι η σωστή λύση για μια σχέση με τους πολίτες. Η σχέση αυτή με τους πολίτες δεν υπάρχει εδώ και χρόνια. Πρόεδρος. Βέβαια έφυγε ο κύριος Ρωμάνο. Θα του μεταφέρουμε τους λόγους σας με τα γραπτά πρασεκτικά. Έχει δεσμευτεί να δώσει συγκεκριμένη απάντηση. Θα δώσει και στην τελευταία ομιλία. Και ίσως και λεπτομέρειες για αυτά που είπατε. Πιστεύω ότι πολλά από όσα υπόθηκαν σήμερα τα σημείωσαν οι συνάδελφοι, θα μπορούσαν ενδεχομένω να μετατρέψουν σε τροπολογίες και το Σεπτέμβριο να μπουν σε ένα κείμενο που θα ψηφίσουμε τέλος Σεπτεμβρίου και θα το στείλουμε στην Κομισιόν. θα ζητήσω μια γραπτή έκθεση επιπλέον της Κομισιόν. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η άποψή σας της Κομισιόν σε σχέση με αυτά που εμείς είδαμε επί τόπου, πώς έχουν τα πράγματα, γιατί αυτό που έγινε ή δεν έγινε στο παρελθόν είτε το θέλουμε είτε όχι, αποκριστελώνεται σε μια απόφαση η οποία εντοπίζει τα λάθη, τις παραβιάσεις, παραβάσεις μάλλον. Βέβαια, όταν υπάρχει δικαστική απόφαση δεν μπορούμε να παρεύουμε. Εμείς ξεκινάμε από την απόφαση του δικαστηρίου και κινούμαστε από εκεί και πέρα. Θα ζητήσω λοιπόν και άλλε διευκρινήσει από την Κομισιόν. Γι' αυτό σα είπα να μα στείλετε ένα γραπτό σημείωμα. Μέχρι τέλο Οκτωβρίου. Α περάσουμε στο επόμενο σημείο. Παρακαλώ του συναδέλφους να κάνουμε μια αντιστροφή γιατί ο χρόνος τρέχει. Είχαμε το 16 αλλά δεν έχουμε κανένα παρόντα αναφέροντα. Γι' αυτό θα δώσουμε ένα πλεονέκτημα στους παρόντες. Δεκαεφτά. Ερμάντο Μενέλα, εκ μέρους της Φέντεραλ Γκίζολε Μινόρι. του δίνω το λόγο να προσθέσει κυρίως νέα στοιχεία αν υπάρχουν. Το θέμα το ξέρουμε. Αν υπάρχουν νέα στοιχεία είτε για την Κομισιόν είτε για μας. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας για την ευκαιρία που μας δίνετε εκπροσωπούμε ξενοδόχους των μικροτέρων νήσων της Ιταλίας. Γνωρίζουμε και εμείς μια περίοδο οικονομικής κρίσης αυτό τον καιρό και διακυβεύεται και κινδυνεύει όλη μας η δραστηριότητα. Γιατί θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν την ε, εταιρεία Τυρένια, ακτοπλοϊκή. Είναι σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχουμε θέσει υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν πολλές άγονες γραμμές. Αν η εταιρεία ιδιωτικοποιηθεί, θα τις καταργήσει. Μαρέτημα, Πόντζα, Λίζο Λαντελζίγιο. Αυτές δεν είναι κερδοφόρες οι γραμμές εκτοπλογικές. Γι' αυτό ζητούμε συμπληρωματικά μέτρα επιπλέον από την αρχή ανταγωνισμού της Ιταλικής Δημοκρατίας για τις ε, εκτοπλογικές υπηρεσίες στον κόλπο της Νάπολης. Βλέπε άρθρο 81 του, της Συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ανταγωνισμού. Θα ήθελα λοιπόν να υποβάλλω ε, στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή τα διάφορα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν γίνεται σοβαστό το άρθρο 81. Στις 11 Μαΐου του 2010 μας απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα έλεγα ότι απορρίπτει ουσιαστικά όλες μας τις ανησυχίες και τα μελήματα, αλλά μας λέει στο τελευταίο τμήμα της απάντησης κάτι σημαντικό. Στα πλαίσια του συμβασμού του κοινοτικού δικαίου, τα κράτη-μέλη έχουν κάθε αρμοδιότητα για να εγγυώνται την εδαφική του συνοχή. Απευθύνομαι λοιπόν στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή και λέγω ότι το Ιταλικό κράτος και οι περιφέρειες είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν την εδαφική αικαιρεότητα. Ευχαριστώ, εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα περιοριστώ κυρίως ε, στα όσα είπε ο προλαλής σας. Για να απαντήσω. Η παρούσα αναφορά αφορά μια κοινοφελή υπηρεσία που είναι οι ε, ναυτιλιακές μεταφορές ε, προς τα μικρά Ιταλικά νησιά. Αυτή η αναφορά ζητεί κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει για να αποφύγει την ε, ιδιωτικοποίηση αυτής της εταιρείας που είναι αυτή τη στιγμή δημόσια και παρέχει μια δημόσια υπηρεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως παρατηρεί το εξής. Τα κράτη-μέλη έχουν κάθε ελευθερία να ε, οργανώνουν τις υπηρεσίες τους με τον τρόπο που θεωρούν σκόπιμο. Και εδώ μιλώ κυρίως για τις ναυτιλιακές μεταφορές, τις αλάσιες μεταφορές. Αν θεωρεί ένα κράτος ότι για ένα νησί θα πρέπει να υπάρχει ένα δρομολόγιο καθημερινό ή θα πρέπει να έχει υπερταχαία πλοία ή με κάποια μορφή ε, αν εσείς ιδιαίτερη στο ταξίδι μπορεί να το κάνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα. Εγώ δεν θέλω να απογοητεύσω τον ε, αναφερόμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να υποχρεώσει το κράτος μέλος να ε, διασφαλίζεται από δημόσιο φορέα η θαλάσσια αυτή μεταφορά. Μπορεί κάλλιστα να οργανώσει τον τρόπο με τον οποίο θέλει το κράτο αυτή την υπηρεσία. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι θα είναι δημόσια υπηρεσία. Δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνε στο κοινοτικό δίκαιο σήμερα είναι ελευθερία του κράτους μέλους και προς τις δύο κατευθύνσεις και στη διοργάνωση της υπηρεσίας και στο να παρέχει ή να μην παρέχει την υπηρεσία αυτή. Αντίθετα, το κοινοτικό δίκαιο τη ζητεί και προβλέπεται και από την αναφορά. Είναι η κοινοφελής αυτή υπηρεσία να παρέχεται εντός του σεβασμού του δικαίου του ανταγωνισμού. Δηλαδή, μια δημόσια εταιρεία ή μια ιδιωτική, μάλλον μια εταιρεία την οποία θα επιλέγει το κράτος μέλος, θα ε, επιλέγεται με μορφή ε, ανταγωνισμού, δηλαδή ε, με δημοπρασία ενδεχομένως, με διαγωνισμό για να υπάρχει ισότητα πρόσβασης στους διαφόρους φορείς που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Για το καμποτάζ που είναι οι θαλάσσιες μεταφορές, Εάν δεν υπάρχει επάρκεια στην αγορά συνδέσεων, το κράτος μέλος στέλνει μάλλον προκυρήσει διαγωνισμό για να επιλέξει την εταιρεία που με το χαμηλότερο κόστος παρέχει την καλύτερη υπηρεσία. Ή όχι και με το μικρότερο κόστος, με το κόστος που ανταποκρίνεται στους πόρους που διαθέτει το κράτος. Λοιπόν, φοβούμε δυστυχώς διαβάζοντας αυτή την αναφορά ότι ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμβαση ε, για το πώς οργανώνει η Ιταλία τις θαλάσσιες μεταφορές της. Μα αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Ούτε έχουμε αρμοδιότητα να αποφύγουμε την απελευθέρωση. Και λυπούμε ότι δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν παρεμβαίνει γιατί δεν είναι δουλειά της. Η πρόεδρο αν μου επιτρέπετε να κάνω μερικέ ερωτήσει στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρατηρήσει γιατί υπάρχουν κάποια σημεία φύση. Διάβασα το κείμενο που μας έστειλε η Κομισιόν, αλλά το θυμήθηκα τώρα που μίλησε ο εκπρόσωπος. Δεν ξέρω αν η αναφορά είναι ασαφής. Εμένα η εντύπωσή μου ήταν διαφορετική σχετικά με, τις, με το αίτημα του αναφέροντος. Ζητάει από την Κομισιόν να ρυθμίσει τις μεταφορές μέσα σε ένα κράτος μέρος. Όχι, ζητάει από την Κομισιόν αν η μέθοδος ρύθμισης της ε, υπηρεσίας μεταφορών, των ουσιαστικών μεταφορών, που σκοπεύει να εισάγει η Ιταλία με την ιδιωτικοποίηση αυτή ανταποκρίνεται στους κανόνες που ορίζει η Ευρωσία με βάση τους όρους συνοχής, άρα προστασίας των πολιτών που ζουν στα περιθώρια και σε δυσμενείς συνθήκες γεωγραφικά. Γιατί και στην Περιφερειακή Επιτροπή ασχολούμαστε με αυτό. Τις προάλλες συζητήσαμε μία γνωμοδότηση εκεί όπου ζητάμε από την Κομισιόν στα πλαίσια της, ε, του καθορισμού της θαλάσσιας πολιτικής να προσέξει κυρίως την ανάγκη τήρησης και σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών που βρίσκονται σε δυσμενείς συνθήκες, άρα να επιμένει η κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων, είτε να ληφθεί υπόψη όσο πρέπει στην πολιτική της εσωτερικής αγοράς, άρα υπάρχει σημαντική αρμοδιότητα της Κομισιόν, και να προωθηθεί η θελάσσια μεταφορά βραχαίων αποστάσεων και το καμποτάζ με καλύτερη σύνδεση μεταξύ περιφερειακών περιοχών και νησιών. Αυτό που συζητάει η Περιφερειακή Επιτροπή είναι ένα κείμενο το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Μια άλλη διευκρίνηση τώρα. Λέτε ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες του κοινωτικού δικαίου. Από την άλλη μεριά, στο έγγραφο που μας διάσατε, μιλάτε για παρέμβαση της Κομισιόν που θα κινήσει διαδικασία παράβασης δεν ξέρετε πού θα καταλήγει, πού θα καταλήξει. Γιατί μια δράση της Ιταλίας σχετική με το θέμα αυτό δεν σεβάστηκε την κοινωτική νομοθεσία, τουλάχιστον αυτό τίθεται ως υπόθεση. Και τέλος. Η Κομισιόν μιλάει μια, μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης που καταρχήν συμφωνεί με τους κανόνες που προσπαθεί να επιβάλλει η έννοια σε όλες τις χώρες μέσω της απελευθέρωσης που ωστόσο ακόμα δεν εγκρίθηκε εκ μέρους της Κομισιόν. Επιφυλάσσεται να κάνει οποιαδήποτε αξιολόγηση ανάλογα με τα πορίσματα της μελέτης των πράξεων σχετικά με τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης στην Ιταλία. Αντιφάσεις αυτά στο κείμενό σας και ανάμεσα στο κείμενό σας και σε αυτά που μας είπατε. Είπατε καμία αρμοδιότητα της Κομισιόν. Η Επιτροπή μας όμως διαπιστώνει ότι τίθεται εν κινδύνο το θεμελιώδες δικαίωμα Ευρωπαίων πολιτών να έχουν την εγγύηση της κινητικότητας που είναι δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη. Η Κομισιόν δεν μπορεί να μην ενδιαφερθεί γι' αυτό, λέγοντας ότι είναι μία αποδεκτή αυτή η αναφορά. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε τώρα ή να μας στείλετε ένα γραπτό κείμενο. Έχετε το λόγο. Μερικές διευθυνήσεις τεχνικές. Το αίτημα ελέγχου συμμόρφωσης της ε, ιδιωτικοποίησης αυτής σε σχέση με την προστασία της ε, ανάγκης κινητικότητας των επιβατών για μας δεν έχει βάση. Δεν υπάρχουν ε, κοινωτικό δίκαιο για την ελάχιστη κινητικότητα των ε, επιβατών. Δύο λόγια. Ένα κράτος μέλος μπορούσε να πει, όσο παράδειγμα και να φαίνεται αυτό, εγώ δεν διασφαλίζω ούτε καν την ελάχιστη υπηρεσία για ένα νησί. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. έχουμε καταγγελίες όταν οι δημόσιες υπηρεσίες παρεμβαίνει, παρεμβαίνουν στο θέμα της απελευθέρωσης της αγοράς. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που δεν αποτελούν παράβαση του κοινωτικού δικαίου. Αντίθετα, το κοινωτικό δίκαιο έχει ένα κανονισμό και γενικές αρχές για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ιδιαίτερα υπηρεσιών και θαλάσσιων μεταφορών. Επειδή η Ιταλία δεν τήρησε αυτούς τους κανόνες, γι' αυτό η Κομισιόν ξεκίνησε μια ανάκριση. Δεν είμαστε ακόμα στη φάση ε, διαδικασίας παράβασης. Στο τέλος του 2008 έληξαν τα δημόσια συμβόλαια της ομάδας της τη Τιρένια και η Κομισιόν περίμενε του επόμενου μήνε να δημοπρατηθούν οι γραμμέ. Δεν έγινε. Ίσως καταλήξουμε σε αιτιολογική σκέψη, κινηθεί δηλαδή η διαδικασία παράβασης. Αν μέχρι το 2010 το τέλος οι Ιταλικές αρχές, όπως υποσχέθηκαν, δεν ολοκληρώσουν το διαγωνισμό αυτό. Η παρέμβαση της Κομισιόν όσον αφορά το κοινωνικό δίκαιο περιορίζεται σε αυτό μόνο. Καταλαβαίνω το πολιτικό σας αίτημα για την πολιτική μεταφορών που θα έπρεπε να ενδιαφέρεται περισσότερο για το θέμα αυτό. Μέχρι στιγμή όμως αυτό το θέμα δεν τίθεται. Σύμφωνοι. Πιστεύω ότι έχετε όμως μια υποχρέωση και αυτή είναι να σέβεστε τις κοινοφελείς υπηρεσίες, τις ελάχιστες. Αυτό αναφέρεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες. Είναι μια υποχρέωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέτε ότι δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα. Ε, τότε Αναρωτιέμαι, τον ξέρετε πραγματικά τον κοινοτικό κανονισμό, τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Σίγουρα είμαστε ένα πολιτικό όργανο, οπότε πιστεύω ότι πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξέρουμε κατά πόσο το τμήμα αυτό τη οδηγία για τις υπηρεσίες έχει απαλληφθεί ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι η οδηγία προβλέπει την εξασφάλιση μια ελάχιστη κοινοφελού υπηρεσία. Όταν μου λέτε ότι ένα κράτο μέλο έχει το δικαίωμα να βγάλει τη σύνδεση μεταξύ κάποιων σημείων της επικράτειας, μου λέτε κάτι ανήκουστο. Ειλικρινά, έτσι όπως γνωρίζω εγώ τα πράγματα, τα κοινοτικά κείμενα, τις οδηγίες, δεν με πείθετε με την απάντησή σας. Συνεπώς, πιστεύω ότι η αναφορά αυτή πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και θα συνεχίσουμε την εξέτασή της στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Ζητάω από τον αναφέροντα. Θέλει και πάλι το λόγο, παρακαλώ. Κοιτάξτε, λέει ο αναφερόμενο, δεν είμαστε κατά της ελευθέρωσης... δεν είμαστε κατά της ιδιωτικοποίηση, εφόσον και εμεί είμαστε ιδιωτικοί φορεί. Θέλουμε όμω να διασφαλίζεται η σύνδεση και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα Ιταλικά νησιά, ισχύει και για άλλα μικρά νησιά. Πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη εξυπηρέτηση σύνδεση. Η Κομισιόν παρενέβη σε άλλες περιπτώσεις και πέτυχε την καταδίκη του Ιταλικού κράτους που είχε μειώσει τις υπηρεσίες αυτές υπερβολικά. Αν καθυστερούμε τη γραμμή Νάπολη-Κάπρη, ε, υπήρχε ανταγωνισμός πριν, υπήρχαν πολλοί φορείς για αυτή τη γραμμή. Σήμερα ένας μόνο φορέα εξασφαλίζει αυτή τη σύνδεση. Ο νόμος του ανταγωνισμού τηρείται, δεν νομίζω. Πρόεδρος. Καλώς, ευχαριστούμε. Ο αναφερόμενο. Ε, μπορώ να δώσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ τα έγγραφα που έχω μαζί μου και που έρχονται από τις αρχές εγγύησης. Εγώ έχω την αίσθηση ότι οι Ιταλικές αρχές δεν τηρούν πάντως τη συνθήκη. Πρόεδρος, θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, να εξετάζουμε την περίπτωση αυτή το Σεπτέμβριο και ενδεχομένως θα προβλέψουμε και μία προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ και περνάμε στο επόμενο θέμα. Πρόκειται για την αναφορά στο σημείο 18. Ιρλανδική ηθαγένεια. Ο κύριος Τζον Μάξ είναι εδώ παρόν, εκ μέρου τη οργάνωση «Οι φίλοι του Λιμένο Πέντζαντ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε από την Κορνουαλή. Σας φέρνω χαιρετισμού. Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να έρθω και να σας μιλήσω για την αναφορά αυτή. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Έρχομαι από το Πενζάνς. Έχουμε 20.000 κατοίκους, είναι στο τέλος της Κορνουάλης, μια πολύ όμορφη πόλη με ιστορικούς χώρους, με ωραία κτίρια και ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. 6.000 τουρίστες έρχονται κάθε χρόνο αλλά είμαστε βέβαια και εργατικό χώρος. Όλα αυτά απειλούνται όμως, διότι θέλει το Συμβούλιο να, χρησι... χρησιμοποιήσει χρήματα για να το κάνει η βιομηχανική ζώνη μέσα σε αυτήν την ιστορική περιοχή. Θέλει να βελτιώσει έτσι το λιμάνι, αλλά αυτό που κάνει είναι ότι επειδή εκεί για να επιτρέψει σε ferry να έρχονται. Αν γίνουν αυτές οι αλλαγές, τότε θα αλλάξει το τοπίο και θα γεμίσει από τσιμέντο ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια της πόλης αυτής που είναι ένας ιστορικός χώρος, ιστορική αποβάθρα και θα κοπεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του ιστορικού χώρου στην πόλη αυτή. Το έργο αυτό θα καταστρέψει τα βικτοριανά κτίρια, τα κτίρια αρντεκό και θα καταστραφούν ε, ακόμα και πουλιά και άλλη πανίδα στην περιοχή. Μας είπαν ότι το σχέδιο αυτό θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης στο Πενζάνς. Όμως εμείς πιστεύουμε ότι θα γίνει ακριβώ το αντίθετο, γιατί οι βελτιώσεις αυτές στο λιμάνι δεν θα φέρουν περισσότερους επιβάτες, Αντίθετα, θα χαθούν θέσει απασχόληση. Προτείνεται να φέρει με μια ενιαία δομή που τελικά θα βολέψει μάλλον τον ιδιωτικό φορέα που έχει αναλάβει το σχέδιο. Το νέο φέρι θα είναι πολύ μεγάλο και έτσι καλώς δεν θα μπορεί να επισκευάζεται εκεί, πράγμα που σημαίνει ότι οι δουλειές σήμερα που είναι για την επισκευή σκαφών θα χαθούν. Τέλος, όσον αφορά τον τουρισμό, θα καταστραφεί ο τουρισμός γιατί θα καταστραφεί το τοπίο. Σήμερα γίνονται διαβουλεύσεις με το τοπικό συμβούλιο που δείχνουν ότι ο χώρος εκεί και το τοπίο είναι πολύ βασικό για την πόλη, ενώ το σχέδιο θα έχει σαν αποτέλεσμα να γεμίσει με φορτηγά και θα καταστραφεί αυτό το ωραίο τοπίο. Μας λένε επίσης ότι ε, τελικά και τα φέρει θα πρέπει να εγκαστούν να πάνε σε ένα άλλο λιμάνι όσο γίνονται τα έργα πάνε στον ιδιωτικό τομέα από το Πεντζάς που ήταν τα τελευταία χρόνια. Και όλοι, ακόμη και ο τρέχον φορέας και το Δημοτικό Συμβούλιο λέει ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί αλλού. Γιατί είναι 40 χιλιόμετρα μακριά το πιο κοντινό λιμάνι, πολύ μακριά από τα νησιά τα οποία εξυπηρετεί. Και θα κοστίζει πολύ χρήματα αυτή η αλλαγή έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θέλουν να πάνε πουθενά άλλου παρά μόνο στο Πενζάνς ε, τα ferry boat που κάνουν τη σύνδεση σήμερα. Οπότε το επιχείρημα του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης δεν ισχύει. Μάλλον θα χαθούν. Έπειτα, οι διευκολύνσεις που έχουμε στο λιμάνι όντω χρειάζονται βελτίωση και θα μπορούσε να γίνει αυτή η βελτίωση με διαφορετικό τρόπο. Και ο κόσμο το θέλει αυτό. Όμω το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διαφορετική προσέγγιση. Εναλλακτικέ λύσει έχουν προταθεί ώστε να προστατευτεί το τοπίο, η υποβάθρα και να προστατευτούν και οι ανάγκε των κατοίκων. Δεν θα γίνει όμω αυτό με ένα fast ferry και με τι αλλαγέ ε, αυτέ που προβλέπονται. Ή δεν έχει γίνει καμιά καλή έρευνα επιμένει το Δημοτικό Συμβούλιο στη δικιά του προτίμησή του και κοφαίνει σε άλλες προτάσεις εναλλακτικέ που γίνονται. Πρόσφατα μάλιστα μάθαμε ότι μια υπηρεσία ελικοπτερού από το Πεντζάν στα νησιά θα κλείσει μέσα στα επόμενα χρόνια γιατί έχουν παλιώσει τα ελικόπτερα και χρειάζονται πολλά καύσιμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο το έχει αγνοήσει αυτό. Ενώ θα υπάρχει το fast ferry για να καλύψει το κενό που θα αφήσουν τα ελικόπτερα δεν προτείνεται ένα νέο σχέδιο με άλλα που θα μπορούσαν να ανακαλύψουν το κενό των ε, ελικοπτέρων αυτών. Η όλη διαδικασία λαμβάνει η χώρα μας λένε βάση των κανονισμών. Δεν είναι αλήθεια όμως αυτό. Η διαδικασία δεν είναι δημοκρατική μας αρνήθηκαν την προστασία που προβλέπεται κανονικά από τις ρυθμίσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο είπε στο κοινό ότι θα έχει την ευκαιρία αν έχει αντιρρήσεις να το πει για το σχέδιο. Στο μεταξύ όμως έχει δυσφαλιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση η αναθεώρηση και μετά μας λένε ότι δεν χρειάζεται να περάσουμε από την συνήθη διαδικασία. Από τη στιγμή που δημοσιεύθηκαν τα σχέδια, ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί κατά του σχεδίου αυτού. Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις εκλογές κανένας δεν το υποστήριξε. Ακόμα και στο Westminster υπάρχουν πολλοί που είναι κατά. Και οι σύμβουλοι για τα παλιά κτίρια επίσης εκφράζουν αμφιβολίες τους για το νέο αυτό σχέδιο. Είμαστε σε δύσκολη οικονομική συγκυρία. Θα έπρεπε να δοθούν χρήματα για άλλα σχέδια και όχι για αυτό το τεράστιο. Οι υπεύθυνοι λένε ότι δεν προσπαθούν να μειώσουν το κόστος στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί τελικά τα χρήματα θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνοι, θέλουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτά πρέπει να δαπανώνται με σωστό τρόπο και για καλό σκοπό. Βοηθήστε μας λοιπόν να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την πόλη μας και τα κοινοτικά κονδύλια να χρησιμοποιηθούν για πράγματα τα οποία χρειάζονται στην περιοχή και στηρίζουν τον κόσμο εκεί. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο εκπρόσωπος Δόκτωρ Δελάγκε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να απαντήσω δίνοντας θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, είναι η σύνδεση των ίσων ΣΥΛΗ με την ε, η Πυρωτική Βρετανία. Και η αναφορά αφορά και, τους, ε, και τις δύο πλευρές, έτσι και τα δύο λιμάνια, ε, Μένω το έργο αφορά και τα δύο λιμάνια, ενώ η αναφορά μόνο το Πενζάνς. Είναι από το πρόγραμμα ΦΕΝΤΕΡ για τη σύγκληση και τη συνοχή. Η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα για το λόγο ότι, όπως γνωρίζει πολύ καλά ο αναφερομένος, δεν έχει εγκριθεί ακόμα το σχέδιο και δεν υπάρχει και μεγάλη ομοφωνία. Θα ήθελα να σας διαβάσω το κανονισμό για τα διορθωτικά ταμεία που ενέκρινε και το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο. Προβλέπετε ότι η διαχειριστική αρχή εκεί, που είναι η αρχή που ορίζουν τα κράτη-μέλη, είναι αρμόδια για την εφαρμογή των ε, προγραμμάτων στα διορθωτικά ταμεία. Δηλαδή, η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να βεβαιωθεί με βάση τον κανονισμό αυτό ότι επιλέγονται τα έργα με κριτήρια που συμφωνίζει η Επιτροπή και δεύτερον, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι ε, είναι συμβατή με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι βασικές αρχές που ε, επικράτησα και τις ε, συνοψίζω, έχουν να κάνουν με τους στόχους των έργων που θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί οι συγκεκριμένοι στόχοι, να αποδεικνύουν ότι είναι απαραίτητα κονδύλια αυτά, ότι υπάρχει σχέση θα πιάσουν ε, τόπο και είναι το κατώτατο απαραίτητο ποσό και επίσης ε, υπάρχει και ένα στοιχείο εφορίας και βιωσιμότητας οποιασδήποτε επένδυσης εκεί. Η διαχειριστική αρχή ε, με την οποία είμαστε σε στενή επαφή ε, ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, συνάδει με τα κριτήρια το πρόγραμμα αυτό και μας ε, αναφέρουν και μερικές ανακτικές λύσεις που έχουν συναναλυθεί. Και επαναλαμβάνω αυτό είναι συμπέρασμα της Εθνικής Διαχειριστικής Αρχής που φέρει την ευθύνη το συμπέρασμα είναι ότι η καλύτερη λύση είναι αυτή που προτείνεται και το καλύτερο δυναμικό για εφορία και βιωσιμότητα για τη διασύνδεση των νησιών Σίλη με την Κορνουάλη. Θα ήθελα να πω επίση κάτι για την νομοθεσία που εφαρμόζεται εδώ. Το βασικό θέμα που διακυβεύεται και φαίνεται ξεκάθαρα στην αφορά είναι οι αποφάσεις και η σύμφωνη γνώμη για το σχεδιασμό της ε, και αυτό είναι θέμα των ε, αρμοδίων εθνικών αρχών. Επίσης, το κτίριο είναι πολιτιστικής αξίας, ε, listed building, ε, είναι διατηρηταίο ως ε, κληρονομιά πολιτιστική και το κτίριο λοιπόν πολιτιστικής αξίας χρειάζεται ιδιαίτερη άδεια. Έχει δοθεί η οικοδομική άδεια από την αρμόδια αρχή, αλλά όχι για το διατηρηταίο. Επίσης θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με την επικουρικότητα. Η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή δεν ε, μπαίνει στα χωράφια αυτά. Επίσης, προφανώς ζητήσαμε τη διαχειριστική αρχή να μας ενημερώνει για την πορεία των διαδικασιών και μας λέει ότι ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητε διαδικασίες, αυτό μας λέγουν οι αρμόδιε αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου και επίσης τα θέματα που αναφέρει ακριβώς αναφορά για την Επιτροπή αυτή ετέθησαν ε, υπόψη των αρμοδίων αρχών στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν απαντήσει σε όλες τις αρχικές αντιρρήσεις και για λόγους διαφάνειας ζητήσαμε αναφορά, ζητήσαμε μάλλον αντίγραφο της αλληλογραφίας και λέγουμε ότι είναι εύστοχες οι ε, παρατηρήσεις. Βέβαια δεν μπαίνουμε στην ουσία για το αν είναι ικανοποιητικέ γιατί είναι θέμα ιστορικό του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάντως, η διαδικασία επιλογής, ε, α πούμε, επιλεξιμότητα για τα κοινοτικά κονδύλια έχει ακολουθεί σωστά και αρμόδιε αρχέ μας είπαν ότι επίση τηρήθηκε πιστά και η εθνική νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Grazie. Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει το λόγο ο συνάδελφος Τάιλ. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή. Ευχαριστώ και τον κύριο Μάξ που έκανε τον κόπο να έρθει από την Κορνουάλη μέχρι εδώ από αυτήν την τόσο όμορφη κομιτεία. Εγώ θα στηρίξω εδώ τους αναφερόμενους και θα ζητήσω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή, ώστε να την ξαναδούμε. Υπάρχουν ε, τέσσερις νομίζω πολύ καλοί λόγοι γι' αυτό, για να μην είναι ανοιχτή η αναφορά. Πρώτα απ' όλα εξέτασα πολύ προσεκτικά την επιστολή της Επιτροπής του Μαρτίου. Μετά πήρα δύο επιστολές από το Southwest από την Περιφερειακή Κυβέρνηση στις 9 Ιουλίου και από την Περιφερειακή Κυβέρνηση του West Midlands 30 Ιουνίου. Και οι δύο αυτές επιστολές εξηγούν ότι ο φύπουργό περιμένει ακόμα για να πάρει απόφαση για το κατά πόσο θα δώσει την άδεια για αυτό το σχέδιο αποφάσισε μάλιστα να εκδώσει μία δήλωση άρθρου 14 στο Συμβούλιο της Κομιτείας ώστε να μην φτάνει η άδεια που είχε αρχικά δοθεί για να προχωρήσει η διαδικασία. Συνεπώς, τι κάνουμε τώρα. Είναι μια μισοτελειωμένη πρόταση ουσιαστικά. Και δεν υπάρχει και τελική απόφαση. Οπότε, σήμερα θα ήταν πολύ πρόημο να κλείσουμε την αναφορά τη στιγμή που οι ίδιες οι αρχές στην Αγγλία δεν έχουν ακόμα αποφασίσει οριστικά τι θα κάνουν. Δεν μιλάω για την ουσία του ζητήματος, λέω απλώς ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει πώς μπορούμε εμείς λοιπόν να απαντήσουμε στην αναφορά αυτή ικανοποιητικά. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να πάρουμε απόφαση σήμερα, είναι ότι συγχρηματοδοτείται το σχέδιο αυτό από, το, από Ευρωπαϊκά Κονδύλια, από το Περιφερειακό Ταμείο και από την Κομιτεία. Δεν υπάρχει απόφαση η χρηματοδότηση δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο εφόσον έχει δοθεί άδεια για το σχέδιο. Γι' αυτό και δεν έχει αποφασίσει ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να άλλος ένας λόγος που πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να περιμένουμε. Συνεχίζω. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε αίτηση στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για συγχρηματοδότηση, που είναι προϋπόθεση για τα χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Σήμερα είμαστε σε οικονομική κρίση και η αγγλική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει περικοπές και θέλουν να περικόψουν από τις δημόσιες δαπάνες μέχρι 40% των δαπανών αυτών. Οπότε, αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη χρηματοδότηση δεν μπορεί να προχωρήσει το σχέδιο. Τέλος, ακούσαμε τον κύριο Μάξ. για το ότι θα χαθούν θέσεις απασχόλησης αν προχωρήσει η πρόταση αυτή. Για διάφορους λόγους που δεν θα σας πω τώρα και δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω εξάλλου ότι η δημιουργία επιπλέον θέσεων απασχόλησης είναι άλλη μία προϋπόθεση για να δοθούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε σας ζητάω για όλου αυτούς τους λόγους να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και θα δούμε. Δεν μου λένε πότε ακριβώς θα πάρουν την απόφαση οι αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ότι θα την πάρουν αυτή την απόφαση όπου να είναι. Πρόεδρος. Δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει. Θεωρώ και εγώ ότι πρέπει να μείνει ανοιχτό το θέμα. Γιατί η πλήρη απάντηση δεν δόθηκε σε ερωτήσεις ούτε στη γραπτή απάντηση ούτε στην προφορική παρουσίαση της Κομισιόν. Ο υπεύθυνο της Κομισιόν για την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή απάντησε σχετικά με την χορήγηση κονδυλίων είπε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους της Κομισιόν να ελέγχεται τα επιμέρους προγράμματα. Άρα αποκλείει ευθύνη της Κομισιόν. Από την άλλη μεριά έχουμε τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλον που πρέπει να δει από κοντά τα προγράμματα. Αν όχι αυτά που χρηματοδοτεί η Ένωση, θα πρέπει να ελέξει αν είναι σύμφωνα με την ε, νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Μια καταγγελία παράβασης της νομοθεσίας για το περιβάλλον που μεταξύ άλλων χρησιμοποιεί και κοινωτικά κονδύλια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για να δούμε αν τα προγράμματα αυτά συμφωνούν με την οδηγία για το περιβάλλον. Και μετά, αφού έχουμε τα στοιχεία αυτά, θα δούμε τι θα κάνουμε. Παρακαλώ τη Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον να δώσει πιο λεπτομεριακή απάντηση στην αναφορά. Θα την ξαναδούμε το Σεπτέμβριο. Τελειώνουμε εδώ, εξηγήσαμε όλα τα σημεία. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Εύχομαι Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ραντεβού. Α, ο Ντέβιντ μου λέει υπάρχει ένα σημείο. Α, το τμήμα Β, οι αναφορές η 87 ένας συνάδελφος μας είπε ότι έπρεπε να είναι στο τμήμα Α. Οι 54, οι 21 και οι 22 το ίδιο να πάνε στο Α.